Από ό,τι έχω καταλάβει, έχουμε συμφωνήσει για ένα εργαστήριο, έτσι δεν είναι, ή ακρόαση θα κάνουμε στις 15 Απριλίου για το θέμα αυτό. Που βέβαια θα δώσει την ευκαιρία στους σκιώδεις και σε εσά την ίδια να ανταλλάξετε παρετέρω απόψει με ειδικού. Τώρα πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο γιατί στις 10 έχουμε μια ακρόαση και έχουμε και μια παρουσίαση στις 9.30. Οπότε θα ήθελα η κυρία Σαρτόρη πρώτα απ' όλα να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες και μετά να ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές και ό,τι σύντομα σχόλια υπάρχουν να τα ακούσουμε. Μετά έχουμε και την Επιτροπή, ε, τον κύριο Σπέση είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά παρακαλώ να κάνετε πολύ σύντομα σχόλια κι εσείς. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έτσι κι αλλιώς στην ακρόαση θα έχετε περισσότερο την ευκαιρία να μιλήσετε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχουμε διάφορες τροπολογίες. 22 Μαρτίου θα είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών έτσι και αλλιώς, γιατί στην Εμότυπη της Ουσίας ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, είναι τέτοιες οι προθεσμίες που δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη δικιά μας. Λυπάμαι γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ήδη έχουμε ανταλλάξει απόψεις, οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Σαρτόρη να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή που ανταλλάσσουμε απόψεις για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, θα ήθελα κυρίως να, πληροφορήσει την, να πληροφορήσω την Επιτροπή μας εδώ για την εργασία την οποία έχω κάνει μέχρι τώρα. Στις 3 Μαρτίου εστάλει το αίτημα και ο κανονισμός και επομένως εγώ στο προσχέδιό μου έχω λάβει υπόψη αυτό τον κανονισμό ε, βλέποντας τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με την ε, πρόταση κανονισμού ε, όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά αλλά και την χρήση βιοκτώνων. Έχουμε 100 τροπολογίες οι οποίες στόχο έχουν την απλούστευση και την εναρμόνιση των διατάξεων για τα κράτη-μέλη και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν επικαλύψεις ε, σε σχέση με τις διατάξεις ε, για τις χημικές ουσίες ε, καθώς επίσης και οτιδήποτε σχετίζεται με την προστασία των καταναλωτών. Βεβαίως, κύριο μέλημα είναι η προστασία των καταναλωτών στις τροπολογίες, στις, ε, στα άρθρα 25, 28, 29 και άλλα ε, έχουμε συνεργαστεί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τα θέματα τα οποία εγώ έλαβα υπόψη μου βεβαίως έχουν ξεπεράσει τις ε, τροπολογίες τις οποίες υποβάλαμε από κοινού ο στόχος μας είναι κυρίως να μειώσουμε τους χρόνους και επομένως και το κόστος που σχετίζονται με την καταχώρηση και αξιολόγηση των ετοιμάτων. Αυτή η δέσμη τροπολογιών από την τροπολογία 18 μέχρι την 62, 18, 19, 20, 22, 50, 60, 61, 62, έχουν ακριβώς αυτό το στόχο, μείωση χρόνων και, και κόστους. Υπάρχουν μετά πέντε τροπολογίες ε, οι οποίες αφορούν καλύτερο ορισμό των διοικητικών τροποποιήσεων ε, αδειοδότησης. Μια τρίτη ομάδα αφορά την βελτίωση των ε, δραστηριοτήτων αλλά και των απαιτήσεων πρόσβασης ε, στα δεδομένα έτσι ώστε ε, να υπάρξει καλύτερη διευθέτηση του φαινομένου free riders, κυρίως μέσω καλύτερου ορισμού του άρθρου 83. η έλλειψη καταχρηστικής διακριτικής μεταχείρισης σε κάποιων προϊόντων που δεν ε, μπορούν να υπαχθούν στην περιγραφή του άρθρου 5, αυτή είναι η τροπολογία 15, ο περιορισμός της ε, ε, συγκριτικής αξιολόγησης για προϊόντα για τα οποία υπάρχει η απαραίτητη εμπειρία καθώς επίσης και η βελτίωση της επισήμανσης με στόχο βεβαίως στην ετικέτα να παραμείνουν μονάχα οι πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για τον καταναλωτή ενώ στο εσωτερικό δηλαδή στα δελτία ασφαλείας θα αναφέρονται οι πληροφορίες οι οποίες δεν είναι άμεσα απαραίτητες καλύτερη ισορροπία για, την το παράλληλο εμπόριο, για, τις, για τα ταυτόσιμα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στις ίδιες δραστικές ουσίες και στο ίδιο περιεχόμενο, βελτίωση των διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αδειών, είναι οι τροπολογίες 52 μέχρι 59, η ευθυγράμμιση των διατάξεων του κανονισμού με την υφιστάμενη νομοθεσία, κυρίως δε με το REACH, με στόχο φυσικά να μην δημιουργηθούν επικαλύψεις. Έχω προτείνει κάποιες τροποποιήσεις έτσι ώστε ε, οι διατάξεις σχετικά με την πρόθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων να είναι απλές, κυρίως ε, για μικρές και μεσαίες βιομηχανίες που αφορούν το 75% ε, των βιομηχανιών που δρούν στην αγορά. Επίσης να υπάρχει ένα ε, κεντρικό, μια κεντρική υπηρεσία ε, η οποία θα ασχολείται με τα ε, αιτήματα διοδότησης όπως προβλέπεται στο Ρίτσο. Τέλος προτείνω την άρση της ετήσιας αξιολόγησης των δασμών προς πληρωμή ε, ε, ε, και οι δασμοί να αφορούν τις εργασίες οι οποίες έχουν πραγματικά λάβει η χώρα. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, είμαι πάντα στη διάθεσή σας να τις συζητήσουμε και αν θέλετε περαιτέρω αποσαφηνήσεις βεβαίως είμαι στη διάθεση των συναδέλφων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την τόσο εξαντλητική εργασία την οποία έχετε κάνει. Είναι πολύ σημαντικά και αυτά τα οποία είπατε σχετικά με τη συμφωνία την οποία επιτύχαμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος στα πλαίσια της ε, συνεργασίας μας και είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για την αμοιβαία αναγνώριση λοιπά. Αυτές είναι τροπολογίες οι οποίες βεβαίως αμέσως θα πάνε στην ε, Ολομέλεια ενδεχομένως ε, θα χρειαστούν αργότερα και κάποιες επιπλέον διαπραγματεύσεις και εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής θα αναμειχθώ προσωπικά στη διαδικασία. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι ε, υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία και αυτό είναι πολύ θετικό. Ε, έχουμε κάποιους σκιώδεις εδώ, ο κύριος Μπορζόη, ο κύριος Φόξο και ο κύριος Βάμπ. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπορζόη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο αυτή την έκθεση, η οποία πραγματικά είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί η πρόταση για τα βιοκτώνα είναι πολύ περίπλοκη και γιατί δεν είναι και εύκολο το θέμα. Οι διαπραγματεύσεις που έκανε η συγκήτρια ήταν πραγματικά αξιέπαινες. Να πω καταρχήν ότι συμφωνώ με τη γενική γραμμή της ε, πρότασης Υπάρχουν ε, αρκετέ ε, ιδέε τι οποίε μπορώ να υποστηρίξω, να δώσω έτσι λίγο έμφαση στη στην διαδικασία αποκεντρωμένη έγκριση που θα μπορέσει να ενισχύσει την ε, αποτελεσματικότητα τη όλη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να προτείνω κάποια επιπλέον στοιχεία, τα οποία θα αποτελέσουν και κομμάτι των τροπολογιών που θα υποβάλω. Καταρχήν, πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία μεταξύ τη προστασία τη ανθρώπινη υγεία και του περιβάλλοντο και του να επιτρέψουμε την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Γιατί πολλέ νέε ουσίε, ε, ο αριθμό των νέων ουσιών είναι πολύ μικρό και γι' αυτό θα ήθελα να, να επιτείνουμε την ε, σημασία τη ε, ανάπτυξη και τη έρευνα και να, έχουμε, και να βασιστούμε και στην πρόταση της Κομισιόν ως προς αυτό για την έγκριση των προϊόντων. Πρέπει να πω ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω μια συγκεκριμένη περίοδου όπου η αρμόδια αρχή μπορεί να εκδώσει μια γνωμοδότηση για τους κινδύνου που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την θέση σε εμπορία αυτού του προϊόντος. Επίσης πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και αυτό μπορούμε να το κάνουμε κάνοντας διαχωρισμού μεταξύ των διαφόρων εγκρίσεων που υπάρχουν στην πρόταση και απλουστεύοντας τι διαδικασίε που είναι σημαντικέ και χωρίς να αυξάνουμε τον κίνδυνο για την ασφάλεια της υγείας και για, τον, για το περιβάλλον. Έχω κάποια σχόλια για τις απαιτήσει ετικητοθεσίας για τα υλικά. Το είχα πει όταν συζητήσαμε τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν οι καταναλωτές. Νομίζω ότι οι πάρα πολλές πληροφορίες τελικά κάνουν ζημιά. Πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που να στοχεύει τον καταναλωτή. Οι απαιτήσει που επιβάλλει η Κομισιόν νομίζω ότι πάνε λίγο μακριά επιβάλλουν, επιβάλλουν ε, άχθος χωρίς λόγο στι επιχειρήσεις και δεν υπάρχει και κανένα, καμιά προσθέμενη αξία για τους καταναλωτές. Και επίσης ε, οι απαιτήσει ε, για την παροχή έγκριση και αριθμού όλων των βιοκτώνων για, το, για, τα, για την επεξεργασία υλικών. Εδώ όμως μιλούμε για τους καταναλωτές οι οποίοι δεν είναι και ειδικοί και θα γίνουν ξαφνικά πιο έμπειροι όταν ξέρουν ποιο είναι το νούμερο αυτών των προϊόντων. Δεν νομίζω. Πρέπει η έκθεση να είναι σαφή, εύληπτη και νομίζω ότι πρέπει να αναλύσουμε και τη δυνατότητα να μπαίνει στην ετικέτα το, το, το όνομα της ενεργού ουσία, χρησιμοποιώντα όμως όπου είναι δυνατόν την κοινή ονοματολογία. Γιατί αλλιώς οι καταναλωτές ε, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μακρύ κατάλογο με άγνωστες ουσίες που ούτω ή άλλω δεν του λένε και τίποτα και πραγματικά καθιστούν την ετικέτα άχρηστη. Και κάποιε άλλε προτάσει έχω, αλλά θα σταματήσω εδώ γιατί δεν συζητούμε τώρα ει βάθο τη τροπολογία. Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι την κυρία Σαρτόρη και ελπίζω στο τέλο να υπάρξει τελικά συνένεση και εδώ αλλά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ελπίζω να μπορέσετε όντως να πάρετε και εσείς σε μέρος uh, στο εργαστήριο αυτό, γιατί είναι καλό η κυρία Σαρτόρη να έχει την υποστήριξη της Επιτροπής στο, um, στο εργαστήριο. Ο κύριος Φόξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Σαρτόρη για την πρόοδο στον, στον ντοσχέ αυτό και για την προσέγγιση που έλαβε. Και με την Ήτρα είμαστε σε στενή ε, συνεργασία και με το περιβάλλον. Θεωρούμε ότι έχουν καλυφθεί σχεδόν όλες οι ανησυχίες μας και Χαίρομαι που θα αποκοινούμε την κυρία Σαρτόρη, θα υποβάλουμε μια τροπολογία ώστε να ε, ε, βελτιωθεί η κεντρική διαδικασία έγκρισης, έτσι ώστε μέσα από αυτό το δρόμο να εγκρίνονται ακόμη περισσότερα προϊόντα. Εγώ με, θα υποβάλω με κάποιους άλλους συναδέλφους κάποιες τροπολογίες για, την, ε, για τις απαιτήσει της έρευνας και της ανάπτυξης, για, για το πεδίο εφαρμογή του του κανονισμού για ουσίες που καλύπτονται και από, την, από τον κανονισμό για, τις, για τα τρόφιμα και επίσης για να βελτιώσουμε το τι θα αναγράφεται πάνω στις ετικέτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σφάμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια και να θυμίσω ότι στην Επιτροπή αυτή έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για χημικές ουσίες και για κανονισμού στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν είχαμε κανέναν από τους πράσινους ή τους σοσιαλιστές, οπότε δεν γινόταν καμιά σοβαρή συζήτηση. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Χαίρομαι που και αυτό έχουμε, γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυρία Σαρτόρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ δεν έχω να υποβάλω οποιαδήποτε τροπολογία, δεν έχω προτιμάσει και ούτε θα προτιμάσω νομίζω ότι δεν είναι, απαραίτητο, Ο στόχος είναι η απλούστευση της όλης διαδικασίας για την αξιολόγηση των ενεργών ουσιών, για, την, για τις χημικές ουσίες και νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνει πρώτα της κυρίας Σαρτόρη. Γιατί πραγματικά έχουμε και το θέμα της εσωτερικής αγοράς και έχουμε μια κατάσταση όπου ε, υπάρχει μεγάλη παρέμβαση των εθνικών πολιτικών. Ε, πρέπει επίσης να επιτύχουμε και την ε, ε, διευκόλυνση σε ό,τι αφορά το διοικητικό άχθος και να δούμε τι γίνεται και με τις ανάγκες ρύθμιση. Επίσης το θετικό είναι ότι σε ό,τι αφορά τα βιοκτώνα δεν πρέπει να μειώσουμε την προστασία των καταναλωτών. Αλλά νομίζω ότι αυτό το επιτυχαίνει η πρόταση τη κυρία Σαρτόρη, οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλοι πήραν το λόγο από τους σοσιαλιστές. Δεν είναι εδώ η κυρία Κέπαρτ. Οπότε, η Επιτροπή τώρα. Ο κύριος Πέτ, θέλετε εσείς να μας πείτε, έχουμε λίγο χρόνο, δώστε μας την αρχική σας εντύπωση επί των τροπολογιών Σαρτόρη και ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την κυρία Σαρτόρη για την επικοδομητική της έκθεση. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία ευχαρίστω να δεχτούμε. Καταρχήν θέλω να πω ότι πολλά από τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε σχέση με την αξιολόγηση και σε σχέση με την μεθοδολογία όπου γίνεται μνήα στα υπάρχοντα δεδομένα είναι πράγματα πολύ θετικά και συμφωνούμε για την ε, σήμανση. Έχουμε πει ότι εμείς θέλουμε μια καλή ισορροπία, οπότε ευχαρίστως να δούμε τις προσεγγίσεις που προτείνει για να έχουμε μια ισορροπία. Για την αηφόρο χρήση των διοκτώνων τώρα. Όπως έχουμε πει και νωρίτερα, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που απαιτεί πολλή δουλειά, αλλά το θέμα είναι η μεθοδολογία στην τροπολογία 28 που αναφέρεται στο δικαίωμα πρωτοβουλίας Οι πιο δύσκολες για μας τροπολογίες, κοιτάξτε, ξέρω ότι ορισμένες θέλουν να περιορίσουν το χρονοδιάγραμμα. Συγχρόνως υπάρχουν και κάποιες άλλες που βάζουν παραπάνω δουλειά, φόρτο εργασίας. Εγώ θα ήθελα να δούμε γενικά τον ε, φόρτο εργασίας και το χρονοδιάγραμμα και όχι κομματάκι-κομματάκι, το σύνολο να είναι λογικό και να μην κάνει τη ζωή δύσκολη στους ενδιαφερόμενους. Όπου έχουμε νούμερα αναφοράς, ε, ρυθμίσεις, ειδικά νούμερα ε, καταγραφής, Αυτά αναρωτιέμαι. Δεν είναι υπερβολικά λεπτομερή γι' αυτό το αρχικό στάδιο ρύθμισης. Μήπως δεν έχει νόημα να τα βάλουμε τώρα και να αναγκαστούμε μετά να τα βγάλουμε. Επίσης για την τροπολογία 24 νομίζω ότι αποδυναμώνει κάπως το στόχο. Όσον αφορά τώρα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Ο λόγος που αλλάξαμε την κατάσταση στην πρότασή μας είναι ότι από την ανάλυση μας ήταν πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε, να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις αυτών των προϊόντων. Γι' αυτό επίτηδες εξαιτία της εμπειρίας που έχουμε μέχρι τώρα για την επεξεργασία τέτοιων ε, προϊόντων, γι' αυτό τα αφήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σαρτόρη τώρα και μετά θέλω να επιβεβαιώσω το χρονοδιάγραμμα, έτσι. Να μας πείτε κι εσείς αν συμφωνείτε, είναι αυτό που περιμένετε. Οπότε, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι 22 Μαρτίου. Ξέρω ότι είναι πολύ σύντομα, αλλά νομίζω ότι οι σκιώδες είναι έτοιμοι γι' αυτό. Έπειτα, να ξαναδούμε τις τροπολογίες της 7 Απριλίου και να ψηφίσουμε πριν από το εργαστήριο. Πριν από τις 8 Απριλίου ή 8 Απριλίου, για να ε, μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα και με το χρονοδιάγραμμα της Επιτεσουσίας Αρμόδιας Επιτροπής. Εντάξει, αν υπάρχουν και συμβιβαστικέ, 7 Απριλίου πρέπει να τις έχουμε. Λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο για να κλείσουμε αυτό το θέμα και για να απαντήσετε σε ό,τι θέματα έθεσαν ενδεχομένω οι σκιώδες συζητητές και η Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς κυρίως γιατί συμβάλατε τα μέγιστα και στην συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και βεβαίως αυτή η συνεργασία συνέβαλε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία ε, την οποία προσπαθούμε να εκπονήσουμε σε σχέση με τον λόγο κανονισμό και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, ε, σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία την οποία είχαμε του τελευταίου μήνε Αναμένω τι τροπολογίε του έτσι ώστε να φτάσουμε σε όσο γίνεται καλύτερε και περισσότερε συμβιβαστικέ λύσει. Ε, και με την Επιτροπή βεβαίω θα έχουμε επαφή έτσι ώστε και η Κομισιόν να κατανοήσει την αιτιολόγηση όλων των ε, ε, τροπολογιών μα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Σορτόρη, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστούμε και την Κομισιόν και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ευτυχή έκβαση ε, όσον αφορά την γνωμοδότηση. Αυτή, ε, όπως είπατε και εσείς, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει με την Επιτροπή, οι επαφές και οι συνεργασίε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Λοιπόν, ε, θα σταματήσουμε τώρα. Θα έχουμε ένα πολύ μικρό, πολύ σύντομο διάλειμμα μέχρι τις 9.30 έτσι ώστε να έρθουν και οι προσκεκλημένοι μας. και νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε όλοι εδώ έτσι ώστε να ακούσουμε ε, την, ε, πολύ, τις πολύ σημαντικές ε, ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ακρόασης και προηγουμένως να ακούσουμε και τον κύριο Τρασόφσκι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμά μας σήμερα το πρωί. για την εσωτερική αγορά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. Λοιπόν, καταρχήν θα μας κάνει μια παρουσίαση η καθηγήτρια Κριστίνα Τόμπλα και θα έχουμε έτσι την παρουσίαση της ως υλικό για την, για την συζήτησή μας. Πρέπει να χρειάζεστε την κάρτα σας. Δεν έχουμε αλλάξει τη θέση σας. Είναι εδώ λοιπόν στο βήμα η κυρία Τόμπλερ για να μας κάνει την ε, παρουσίασή της. Ε, οι εμπειρογνώμονες είναι εδώ μπροστά για την ακρόαση στις, που θα ξεκινήσουμε στις 10. Και χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω και τον εισηγητή μας για την πολύ σημαντική αυτή έκθεση, τον κύριο ε, ο οποίος κάνει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και ως Επιτροπή θεωρήσαμε ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία στην αρχή αυτής της πενταετίας η Επιτροπή μας να καταγράψει ποιες είναι οι σχέσεις μας στην εσωτερική αγορά με τους πολύ σημαντικούς εταίρους μας και τους γειτόνους μας και να συμμετέχουμε όλοι σε αυτή τη διαδικασία της εκπόνησης πολιτικών. Μία από τις βασικές αποστολές της Επιτροπής μας δεν είναι να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία, που εντάξει έχουμε και μια ευθύνη και γι' αυτό, αλλά είναι να ε, αξιολογήσουμε όλο το κεκτημένο για την εσωτερική αγορά, που δουλεύει, που δεν δουλεύει και προς το παρόν έχουμε δύο παράλληλες ε, δουλειές που γίνονται, μία για τις δημόσιες προμήθειες μία για την, και μία για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων. Ε, όπου σκεφτόμαστε το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει μια, μια μεταρρύθμιση και να δούμε πώς γίνεται να μεταφερθεί καλύτερα η ε, οδηγία ας πούμε, για τις υπηρεσίες, ε, το πακέτο για την εποπτεία της αγοράς και τα αγαθά και τα διεθνή πρότυπα το, για, για τα οποία θα υπάρξει μια νομοθετική πρόταση προς το τέλος του χρόνου. Φιλόδοξη λοιπόν η ατζέντα μας και ένα τμήμα αυτής της δουλειάς είναι να φτάσουμε στους εταίρους μας όχι μόνο στον ΕΟΧ και στην Ελβετία, αλλά έχουμε και πάρα πολλέ πολλέ συναντήσεις από διάφορους, από διάφορους βουλευτές, από διάφορα κρατημέλη. Αυτά λοιπόν έτσι εισαγωγικά. Οπότε, προς το παρόν να δούμε την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της καθηγήτριας Τόμπλερ. Είναι καθηγήτρια ε, νομικής στην ε, Βασιλεία και ειδικεύεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο πώς αυτό συνδέεται ε, και με την νομοθεσία που διέπει την Ελβετία και με την νομοθεσία που διέπει τον ΕΟΧ. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Τόμπλερ για να μας κάνει την παρουσίασή της. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομα θα σας αναφέρω ποια είναι τα βασικά σημεία του ενημερωτικού σημειώματος που έχετε μπροστά σας. Το ενημερωτικό αυτό σημείωμα αφορά την εσωτερική αγορά πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή η Κοινή Αγορά ε, διέπεται από ελεύθερη κυκλοφορία ε, κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αυτό συμπληρώνεται από σημαντικούς κανόνες ανταγωνισμού. Το δίκαιο ανταγωνισμού δεν ήταν το επίκεντρο αυτής της μελέτης, ήταν κυρίως οι τέσσερις ελευθερίες. Αυτά ως αρχικά σχόλια. Η μελέτη αυτή έχει να κάνει με την επέκταση της ιστορικής αγοράς πέρα από, τις από, την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ε, υπάρχουν οι κανόνες της ιστορικής αγοράς οι οποίοι όμως ε, αφορούν μόνο και εφαρμόζονται μόνο στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν αυτοί οι κανόνες ή παρόμοιοι έχουν ε, επεκταθεί και σε άλλες χώρες μέσω ε, συμφωνιών και αυτό που κάνει η έκθεση είναι να βλέπει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις από τη μία την, ε, τις χώρες ε, ΕΟΧ και ΖΕΣ και από την άλλη την ε, Ελβετία. Στην επόμενη διαφάνεια. Ο στόχο αυτού του ενημερωτικού σημειώματο είναι να δούμε ποιο είναι το εύρο αυτή τη ιστορική αγορά σε ό,τι αφορά αυτέ τι δύο ομάδε χωρών. Για να δούμε, και το κάνουμε αυτό βλέποντα δύο τελείω διαφορετικά μοντέλα ολοκλήρωση, έτσι ώστε να βρούμε ποιε είναι οι προκλήσει και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την, απόδοση αυτή της ενισχυμένης ε, διευρυμένης εσωτερικής αγοράς. Τα δύο μοντέλα για τα οποία μιλούμε βασίζονται σε αρκετά διαφορετικά νομικά πλαίσια. Το σύστημα ΕΟΧ είναι πολυμερές ε, πλαίσιο που σημαίνει ότι έχει αρκετέ, υπάρχουν αρκετές τρίτες χώρες το, η Ελβετία και το σχετικό μοντέλο είναι διμερές, δηλαδή περιλαμβάνει μόνο την Ελβετία και αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ο αριθμός των, των συμφωνιών που υπάρχουν στα πλαίσια του ΕΟΧ. Υπάρχει μια συμφωνία η οποία βέβαια ρυθμίζει όλο το εύρος των σχέσεων. Ε, στην Ελβετία έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό συμφωνιών, πάνω από 120 σήμερα υπάρχουν, που ε, και αυτό από μόνο του είναι πρόκληση. Και παρόλο που υπάρχουν αυτές οι 120 συμφωνίες, υπάρχουν οι 20 οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος. Οπότε είναι αρκετά διαφορετική η κατάσταση η δική μας. Όταν, αν δείτε το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών, των δύο συστημάτων, θα δείτε ότι έχουμε πραγματικά αρκετά σημαντικό, αρκετά διαφορετικούς βαθμούς του ε, κοινοτικού δικαίου. Ε, για τον ΕΟΧ μπορεί κανείς να πει ότι είναι απλουστευμένος, ότι το σύστημα ας πούμε, ε, είναι συνολικό. Δηλαδή περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν όλα από όσα περιλαμβάνονται στο κοινοτικό δίκαιο. και οι τέσσερι ε, ελευθερίε περιλαμβάνονται εδώ με κάποιες εξαιρέσει. Αν δείτε όμω τον, τον, το άλλο μοντέλο, θα δείτε ότι είναι αρκετά επιλεκτικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και τονίζεται και από το δικαστήριο στην πρόσφατη νομολογία του. Είναι επιλεκτικό λοιπόν σύστημα. Δεν είναι σύστημα που περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν περιλαμβάνει το σύνολο του μοντέλου τη εσωτερική αγορά. Αν δείτε λοιπόν τι τέσσερι ελευθερίε, θα δείτε ότι καλύπτονται κατά μεγάλο βαθμό τα αγαθά, αλλά όχι πλήρω. Αν δείτε τα άτομα, θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλος περιορισμός ε, για την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών. Μιλούμε δηλαδή μόνο για φυσικά πρόσωπα και αυτό σε περιορισμένη βάση. Επίση, οι υπηρεσίες πάρα πολύ, πάρα πολύ κυρίως γιατί δεν έχουμε συνολική συμφωνία για τις ε, υπηρεσίες και έχουμε μεγάλα κενά. Ε, το, τα η ελεύθερη κυκλοφορία και κεφαλαίων δεν καλύπτεται καθόλου. Αν δείτε λοιπόν τα βασικά από τι τέσσερι ελευθερίες, το πρώτο σημαντικό έβριμα είναι ότι το διμερές σύστημα είναι επιλεκτικό σύστημα, παίρνει κάποια ε, κομμάτια τομεακών ε, συμφωνιών όπως τις, λέμε στην Ελβετία και δεν ε, έχει ως στόχο να είναι συλλογικό. Έχει ως στόχο να είναι αυτό που είναι, επιλεκτικό. Επίσης, έχουμε κάποιους περιορισμούς, όχι μόνο στο πεδίο εφαρμογής. Αν δούμε δηλαδή την, το εύρος της εσωτερικής αγοράς, έχουμε και κάποιους περιορισμούς από πλευράς χρόνου. Αν δείτε το σύστημα ΕΟΧ, μπορείτε να το θεωρήσετε ιδιαίτερα δυναμικό είναι αλήθεια ότι βασίζεται στην νομοθεσία ως, ε, ήταν, ως, ως, όταν υπήρχε, όταν υπεγράφησαν οι συμφωνίες, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηλαδή, αλλά έχει σε κάποια σημεία ε, ενημερωθεί ό,τι φορά τη δευτερογενή νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ δυναμικό λοιπόν. Αν δείτε τώρα σε σύγκριση το διμερές δίκαιο, στην, ε, τη διμερή συμφωνία με την Ελβετία, είναι αρκετά στατική βασίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο όπως είχε αυτό όταν υπεγράφησαν οι εν λόγω συμφωνίες ενημερώνεται σε ένα βαθμό γιατί οι μικτές επιτροπές έχουν αρμοδιότητα να τροποποιήσουν κάποια παραρτήματα ή και την ίδια τη συμφωνία σε μερικές περιπτώσεις για να την ενημερώσουν αλλά είναι περιορισμένο, είναι αρκετά περιορισμένο. Και αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι μετά την ένταξη των νέων κρατών μελών το 2004 δηλαδή και το 2007 ε, με τις σχετικές διευρύνσεις η συμφωνία για την ελεύθερη διακίνηση κυκλοφορία ε, πολιτών δεν επεκτάθηκε για να περιλαμβάνει και αυτού. Οπότε εκεί υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα, συγκεκριμένοι περιορισμοί για το πώς εφαρμόζεται η, ελευθερία της, ε, η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών σε αυτά τα άτομα. Τώρα, μιλούμε για την επιορροή αυτών των, τριών, των τρίτων χωρών στην ε, νομοθεσία που αφορά τα δύο αυτά συστήματα. Αν ε, θα δείτε ότι είναι σημαντικό πώς το δευτερογενές δίκαιο υιοθετείται, ποιος μπορεί να το επηρεάσει, ποιος μπορεί να συμμετάσχει, τουλάχιστον στην, ε, στην ε, εκπόνηση των αποφάσεων, αν όχι στη λήψη αυτών, ε, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει αυτό ως κομμάτι στην ε, διευρυμένη ιστορική αγορά. Στην, ε, στην, στο χώρο ΕΟΧ και ΕΖΕΣ, οι χώρε οι σχετικές έχουν τουλάχιστον κάποιες πιθανότητες να συμμετάσχουν στην εκπόνηση των αποφάσεων. Είναι μέλη αρκετών επιτροπών, μπορεί να είναι παρόντες, μπορούν να συζητούν, μπορούν να δώσουν την άποψή του. Αν δείτε πάλι το διμερές σύστημα με την Ελβετία είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχει κανείς σε επίπεδο εκπόνησης ε, αποφάσεων. Τώρα πάμε στην ουσία. Στην ουσία το εσωτερική αγορά. Τι, τι σημαίνει η ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι το σύστημα ΕΟΧ είναι βασισμένο στην αρχή της ομοιογένειας. Δηλαδή το, δίκαιο σημαίνει το ίδιο όπως και το ευρωπαϊκό δίκαιο που έχει εφαρμοστεί και από το δικαστήριο 7 το οποίο ήταν ε, ιδιαίτερα ε, θετικός προς αυτό. Τώρα για, τον, ε, για τη διμερή συμφωνία με την Ελβετία ήταν λίγο δύσκολο να βρούμε όρο για να σας το εξηγήσω. Είπα ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Ξέρουμε ότι για κάποιες συμφωνίες υπάρχουν όντως διαφορετικές ερμηνείες θα βρείτε λεπτομέρειες και στην έκθεση, μπορούμε να δούμε μια τάση που λέει ότι όντω υπάρχουν διαφορετικά συστήματα, όπω σα είπα πιο πριν. Το ΔΕΚ το λέει επίση ότι δεν είναι απόλυτα δίκαιο εσωτερική αγορά, είναι κάτι άλλο, είναι λίγο πιο τομεακή η προσέγγιση και αυτό έχει ε, επίπτωση και στην ερμηνεία. Αυτό που σημαίνει λοιπόν, ή αυτό που θα μπορούσε να συμβαίνει, είναι ότι υπάρχουν κανόνε για την ελεύθερη κυκλοφορία που δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα εντό του συστήματο του ευρωπαϊκού δικαίου και εντό του συστήματο του διμερού δικαίου με την Ελβετία. Ακόμη και αν δείτε το γράμμα ε, τη νομοθεσία, που μπορεί να είναι, πολύ που μπορεί να είναι παρόμοιο. Τι προκύπτει τώρα σε ό,τι αφορά την νομική ασφάλεια. Υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι εκρεμή, είναι ανοιχτά, συζητούνται, δεν έχουν ληφθεί αποφάσει. Σημαντικά ζητήματα τη εσωτερική αγορά, όπω α πούμε το τι σημαίνει ελεύθερη κυκλοφορία, σημαίνει ελευθερία μόνο για, την, για τη μη διάκριση από άλλες ε, χώρες, σημαίνει κυκλοφορία που σημαίνει ελευθερία ε, χωρίς περιορισμό, σημαίνει κάτι άλλο από την ομολογία, δεν ξέρουμε. Τι σημαίνει όταν μιλούμε για υπηρεσίες και για παραλήπτες, έχουν δικαίωμα πρόσβαση στην αγορά, έχουν μόνο δικαίωμα του να είναι παρόντε σε κάποιο άλλο κράτο μέλο για να λάβουν την υπηρεσία. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Η νομοθεσία λοιπόν εκεί είναι λίγο ασαφή. Υπάρχουν κάποια σημεία λοιπόν τα οποία είναι ακόμη ανοιχτά. Τώρα πάμε στη διαχείριση των, δύο συστημάτων για τα οποία σα μιλώ. Μπορείτε να δείτε στην έκθεση ότι για τον ΕΟΧ και τι σχετικέ συμφωνίε, η διαχείριση σε κάποιε περιπτώσει είναι λίγο δίσκαμπτη. Πρέπει να είμαι ειλικρινή όμω ότι δεν, πρέπει να πω ότι δεν είναι ιδιαίτερο δίσκαμπτη. Λειτουργεί αρκετά καλά, αρκετά καλά το σύστημα. Υπάρχουν κάποιε περιπτώσει που μπορεί να πει κανεί ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει χρονικό κενό για να εγκριθεί το δευτερογενέ δίκαιο. Αν δείτε τώρα τι τις, ε, τις διμερεί συμφωνίε, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι ε, τελείω δίσκαμπτο κυρίως γιατί έχουμε τόσες πολλές μικτές συμφωνίες, γιατί δεν έχουμε ε, πολλές συναντήσεις, ε, δεν υπάρχει γενικώ πολλή συνεργασία, πολλή δράση μεταξύ μα. Η επικοινωνία λοιπόν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Η προσαρμοστικότητα η, ε, τον, και η εφαρμογή των Παρατημάτων και τη νομοθεσία θα, θα έπρεπε να είναι καλύτερα. Γι' αυτό δυστυχώ είναι λίγο δύσκολο ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε, διαχειριζόμαστε αυτέ τι συμφωνίε. Τώρα, παρακολούθηση και εφαρμογή. Βλέπετε ότι έχουμε αρκετά διαφορετική κατάσταση εδώ στα δύο συστήματα. Αν πάρετε τον ΕΟΧ και τη σχετική νομοθεσία, για να το πω απλά, τα, λαμβάνουμε τα βασικά στοιχεία τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχουμε ένα σύστημα δύο πυλώνων, έχουμε την Κομισιόν, ε, ε, έχουμε, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ESA από τις χώρες ΕΖΕΣ, έχουμε το ε, δικαστήριο της ΕΦΤΑ, της ΕΖΕΣ, έχουμε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή αντιστοιχίες. Τώρα, για το διμερές δίκαιο, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι, δεν είναι αποτελεσματικό, απλώ λειτουργεί διαφορετικά δεν έχουμε ε, κοινό σύστημα και το ε, πώς, γίνεται η εφαρμογή αποφασίζεται από τις δύο μεριές. Ε, η επιδροή βέβαια τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά μεγάλη. Στο διμερές, ε, το διμερέ δίκαιο ούτω ή άλλω είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού δικαίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελβετία τώρα είναι λίγο πιο περιορισμένο, γιατί η Ελβετία δεν είναι μέλο, κράτο μέλο. Τα δικαστήρια, α πούμε, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ε, τα ελβετικά δικαστήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τι προδικαστικέ αποφάσει. Δεν μπορούν δηλαδή να πάνε στο δικαστήριο και να ζητήσουν βοήθεια με την ερμηνεία της, ε, των συνθήκων ή κάποιου άρθρου. Οπότε υπάρχουν ανισότητες εδώ στην ε, όλη κατάσταση και υπάρχει ο κίνδυνος κάποια πράγματα να παραμείνουν εκρεμή και να υπάρξουν ε, διαφορετικές ερμηνείες κτλ. Τώρα, γενικώ, ποια είναι τα ευρήματα. Πάω λίγο γρήγορα, αλλά εντάξει. Ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε ό,τι αφορά τον ΕΟΧ, αυτό που υπάρχει είναι ότι είναι, χώρος τη εσωτερικής, είναι κομμάτι της εσωτερικής αγοράς. Ο όρο που αναφέρεται στην ε, έκθεση είναι ότι επί της αρχής είναι βασικό κομμάτι της εσωτερική αγοράς. Είναι συνολικός, υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία και εκτός από την ελεύθερη κυκλοφορία υπάρχουν και κάποιες επιπλέον πολιτικέ οι οποίε συμπληρώνουν την ε, παραδοσιακή, τα παραδοσιακά δικαιώματα ελεύθερη κυκλοφορία. Οπότε γενικώ είναι αρκετά περιεκτικό ο νόμο αυτό. Τώρα για το διμερέ δίκαιο με Ελβετία, όπω σα είπα πριν, είναι επιλεκτικό σύστημα. Η έκθεση λέει ότι η Ελβετία ενσωματώνεται όλο και περισσότερο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια τέτοια διαδικασία ώστε να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι τομεί, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι περιοριστικό το σύστημα και αυτό έχει και ω στόχο να είναι Υπάρχουν πολλές ε, συμφωνίες, ε, είναι αρκετά δύσκολη η διαχείρισή τους, είναι περίπλοκο το θέμα και αυτό που λέει επίσης η έκθεση είναι ότι η Ελβετία μπορεί όντως να διστάζει να αναλάβει, να ενσωματώσει όλες αυτές τις επιπλέον συμπληρωματικές πολιτικές που αποτελούν κομμάτι του συστήματος του ΕΟΧ. Τώρα, ποιες είναι οι συστάσεις. Οι συστάσεις που θα βρείτε στην έκθεση είναι ε, αρκετά λίγε προ έκπληξή σα για τον ΕΟΧ. Κοινοποίηση από την Κομισιόν για τι νομοθετικέ προτάσει. Νομίζω ότι μπορείτε να ενημερωθείτε και εσεί βέβαια, χωρί να το λέει αυτό η έκθεση, ούτω ή άλλω, αυτό γίνεται με τα επίσημα έγγραφα. Δεύτερον, καλύτερη συμμετοχή των χωρών ΕΟΧΕΖΕ στην όλη διαδικασία καθορισμού των αποφάσεων και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Και ένα ενδιαφέρον σημείο, το οποίο το είπα και λίγο πιο πριν, είναι η ενημέρωση τη συμφωνία ΕΟΧ της, αυτής καθ' αυτή της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία ε, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά βέβαια είναι αρκετά δύσκολο, ε, αρκετά περίπλοκο ως καθήκον και μεγάλο. Τώρα, για τις διμερείς συμφωνίες και για τις σχετικές συστάσεις. Η έκθεση αναφέρει πολύ περισσότερα. Λογικό, γιατί είναι πιο περίπλοκο το σύστημα, πιο επιλεκτικό. Και θα δείτε ότι το πρώτο σημείο που αναφέρατε στην έκθεση είναι να δημιουργηθεί πολιτική βούληση και ευαισθητοποίηση ε, για την ε, ε, συνεργασία και για την εντατικοποίηση των διμερών σχέσεων. Ξέρετε ότι η Ελβετία είναι περήφανη για την δημοκρατία της. Έχουμε δημοψηφίσματα για κάποια θέματα. Βεβαίως πρέπει να έχουμε ε, υπόψη ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν δυσκολεύουν λίγο τη ζωή μας. Δεν είναι απλώς μόνο η κυβέρνηση που λέει ας προχωρήσουμε με αυτό και γίνεται. Πρέπει να πιστεί και ο λαός για να γίνει κάτι. Οπότε αυτό είναι το πιο, η πιο μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ. Τώρα, άλλε συστάσει βλέπετε εδώ είναι να γίνονται περισσότερε συνεδριάσει, να εμπλέκεται περισσότερο η Ελβετία στην όλη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ε, Σα ανέφερα το κοινό σύστημα εφαρμογή, αλλά αυτό είναι αρκετά σημαντικό ως καθήκον το οποίο δεν μπορεί εύκολα να επιτευχθεί. Εδώ κλείνω την πολύ σύντομη παρουσίασή μου για τα βασικά σημεία όχι επί της ουσίας ε, της έκθεσης, αλλά ποια ήταν τα ευρήματα που θεώρησα εγώ σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι, έχουν άμεση σχέση φυσικά με το θέμα μας. Θέτεται κάποια ζητήματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία με το πάνελ να τα συζητήσουμε. Δεν έχουμε πάντα αυτή την ευκαιρία και αυτό χαιρόμαστε που ήσασταν εδώ και μπορέσαμε και τα συζητήσαμε. Στις 10 επίσημα ξεκινάμε, οπότε ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάποιες αντιδράσεις από τους ευρωβουλευτές, αυτά που είπατε. Δεν ξέρω εκτός αν ο εισηγητής έχει κάτι να πει. Α, αργότερα εσείς θα μας δώσετε την εισαγωγή σας. Καλά, ερωτήσεις τότε, αν υπάρχουν ε, ερωτήσεις για την ε, καθηγήτρια πριν προχωρήσουμε. Και πριν μπούμε στην ακρόαση αυτή καθ' αυτή. Εσείς και τη ΣΒΑΠ, όχι, όχι. Καλά. Ένα ενδιαφέρον θέμα για μένα τουλάχιστον, μια που έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, γιατί ακριβώ στις 10 θα σταματήσουμε, γιατί έχουμε και την τηλεόραση και φυσικά περνάει στον κυβερνοχώρο η σημερινή μας συνεδρίαση μέσω διαδικτύου. Συνεπώς, αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά για μας. Η με την ακρόαση αυτή κατά κάποιο τρόπο υιοθετούμε κάποιες από τις δικές σας τοποθετήσεις. Αυτό πάντως που πιστεύω ότι βοηθάει πολύ τον κόσμο, όπως και εμένα, που δεν μπορώ να πω ότι έχω τόσο φοβερή σχέση με τους ελβετούς εταίρους μας στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, είναι ακριβώς αυτά που λέτε για το πόσο περίπλοκο είναι το σύστημα της διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ μας. Αυτό το σημείωσε όλος ιδιαίτερος και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα να βρούμε έναν τρόπο που να είναι αποδεκτός από την ελβετική παράδοση και τη δημοκρατία. Εμείς οι Βρετανοί βέβαια καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο που να διευκόλυνε τη διαχείριση των λεπτομεριών των σχέσεών μας. Μιλήσατε για γενικές αρχές, ναι, αλλά η εσωτερική αγορά αντιμετωπίζει συνεχώς αλλαγές. Εξελίσσεται συνεχώς αυτές τις αλλαγές. Πώς θα μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε καλύτερα. Η καθηγήτρια, κοιτάξτε, υπήρξαν πολλές συζητήσεις για τη μελλοντική συμφωνία πλαίσιο. Έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, τις εφημερίδες, ο πρέσβης μας φυσικά είναι πολύ περισσότερο σε θέση να σας τα πει όλα αυτά. Πάντως αυτά που διαβάζουμε στα επίσημα έγγραφα και στις εφημερίδες είναι ότι η ελβετική πλευρά θα ήθελε μια συμφωνία πλαίσιο που να πηγαίνει μέχρι την διαχείριση αυτή καθ' αυτή. Όμω από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ακούμε ότι μια τέτοια συμφωνία πλαίσιο πρέπει να αλλάζει και περισσότερο σε βάθος το σύστημα. Δηλαδή όχι μια συγχώνευση επιτροπών έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η διαχείρισή τους. Όχι, θέλει περισσότερο δυναμισμό στο σύστημα Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου αυτόματα να γίνονται οι προσαρμογές. Η ελβετική κυβέρνηση έχει πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Γιατί δεν ευθυγραμμίζεται με την προστασία της κυριαρχίας μας και δεν μπορούμε τότε να αποφασίζουμε πότε θέλουμε να συμμετέχουμε στο σύστημα. Για μας λοιπόν, όντας εκτός των εσωτερικών συζητήσεων, ε, καταλαβαίνετε μας δυσκολεύει. Έχω την αίσθηση ότι εσείς βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα για το τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε με μια συμφωνία πλαίσιο από ότι εμείς. Και μάλιστα δεν ξέρω καν κατά πόσο θα μπορούσαμε να βρούμε κοινοτόπο μεταξύ μας γι' αυτό όσον αφορά το μέλλον. Ωραία. Ναι, δύο λεπτά, δύο λεπτά πριν ξεκινήσει η μετάδοση. Δύο λεπτά μέχρι να ξεκινήσει η μετάδοση λοιπόν. Σε σχέση και με αυτό που είπατε, δύο παρατηρήσεις να κάνω. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την ε, ιδιαίτερος εύληπτη και γενικόλογη έκθεση. Όντω είναι δύσκολο το να δούμε ποια είναι τα θέματα που αφορούν και την Ελβετία και την ευρωπαϊκή αγορά και πραγματικά υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία που είναι άγνωστα μεταξύ των δύο συστημάτων. Να πω όμως, μια που μιλήσατε για γενικά πολιτικά θέματα, μιλάτε για τους κινδύνου σε κάποιο σημείο της έκθεση, που μάλλον μετά θα δούμε και στη λεπτομέρειά τους για τον κίνδυνο λοιπόν των διαφορετικών ερμηνειών και για τους κινδύνους που, αυτή, που επιφέρει μαζί της αυτή η ιδιαίτερη διαχεί, μεταχείριση. Τι λύσεις υπάρχουν όμως ε, ε, για, τις διαφορετικές αυτές, ε, για τους διαφορετικούς αυτούς κινδύνους πέρα από την διμερή συμφωνία. Θα το πάρω αυτό σαν ένα παράδειγμα. Δεν έχουμε βέβαια χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειε, αλλά το πιο γνωστό παράδειγμα είναι όλη η συζήτηση για το Κασίς Δεντιζού. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ερμηνεία της Συμφωνίας για το Ελεύθερο Εμπόριο του 1972, όπου εκεί υπάρχουν αντίστοιχες διατάξεις όπως το κοινοτικό δίκαιο, αλλά η ερμηνεία είναι διαφορετική. Όλη αυτή η ιστορία της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το Κασίς Dijon» δεν, ε, είναι, δεν έχει την ίδια ερμηνεία στην Ελβετία. Αυτό είναι ένα κατάφορο παράδειγμα. Και μπορούμε να έχουμε προβλήματα και με άλλες συμφωνίες για τους λόγους ε, ακριβώς που έθιξα. Συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε χρόνο, οπότε θέλω να τηρήσω τα όσα ζήτησε ο Πρόεδρος, να πειθαρχήσω. Μα θα έχουμε την ευκαιρία, λέει ο Πρόεδρος, να το συζητήσουμε και στο πάνελ ε, σε λίγο. Έτσι καλώς χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε και τον Ελβετό πρέσβη μαζί μας. Συνεπώς, ε, κλείνει η παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρουσιάσατε το θέμα αυτό. Τώρα θα πάτε με τους εμπειρογνώμονες. Η Αντιπρόεδρος Κορχόλα έφτασε. Καλώς ήρθατε. Εδώ λοιπόν κλείνει αυτό το τμήμα της συζήτησης. Και τώρα μπορούμε να μπούμε στην ακρόαση. Ξεκινάει η ακρόαση. Έχετε, φαντάζομαι, τα έγγραφα στη διάθεσή σας. Υπάρχουν οι διαφάνειες, υπάρχει ένα βιογραφικό των ομιλητών, κάποιες από τις παρουσιάσεις. Τα έχετε αυτά. Συνεπώς, σας καλωσορίζω όλους εδώ. Ευρωβουλευτές, εμπειρογνώμονες, επισκέπτες και το κοινό που μας παρακολουθεί μέσω διαδικτύου, που συντονίστηκε μόλις τώρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και εσείς στη συνεδρία αυτή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εδώ έχουμε μία ακρόαση σήμερα όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. Εμπόδιο όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Θα εξετάσουμε μεταξύ άλλων και τις επιπτώσεις που έχουν οι κοινοτικές ρυθμίσεις στις ε, σχέσεις μας με ζωτικούς για μας ε, εταίρους από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, αν κοιτάξει κανείς τα στατιστικά δεδομένα από το βαθμολόγιο που έχουμε για τις επιδόσεις των χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας, θα διαπιστώσετε ότι κυρίως η Νορβηγία βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στο εθνικό τους ε, δίκαιο. Πολλές φορές ρωτάμε τους πολιτικούς σε διάφορες χώρες εσείς τα πάτε καλύτερα από άλλους. Ε, λοιπόν, να, μια χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία περισσότερα κομμάτια του κοινοτικού δικαίου από ότι χώρες που είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή λοιπόν σκέφτηκε, η Επιτροπή μας, ότι θα ήταν πολύ καλό να έχουμε αυτή την ακρόση. Ο κύριος ε, Τσρασκόφσκι έχει αναλάβει έκθεση από πλευρά της δικιάς μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την πρόταση της Κομισιόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για το ότι ανέλαβε να ηγηθεί και τις ακρόασης αυτής. Οπότε τον καλό να κηρύξει την έναρξη της ακρόασής μας με κάποιες ιδέες, με κάποια θέματα, τα οποία θα ήθελε να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της ακρόασης αυτής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Τρασκόφσκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με ευχαριστίες. Ευχαριστίες προς όλους όσοι έχουν έρθει εδώ, το καθηγητή Τόρτμαν για την εξαίρετη δουλειά εδώ που ετοίμασε το έγγραφο αυτό και θέλω να πω και δύο λόγια για το πλαίσιο και να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Βλέπετε, εμεί αποφασίσαμε να έχουμε καταρχήν ένα έγγραφο εργασία, προκειμένου να μιλήσουμε για τα πιο κέρια ζητήματα. Και είναι ένα έγγραφο εργασία το οποίο μας βοηθάει να εντοπίσουμε κάποια σημεία προς και να τα διευκρινίσουμε. Τελικά όμως θα καταλήξουμε σε μία έκθεση, μετά την ακρόαση βέβαια, γιατί θέλουμε πρώτα να ακούσουμε τι έχετε κι εσείς να μας πείτε, να σκαλίσουμε δηλαδή περισσότερο σε βάθος το θέμα και μετά, αφού έχουμε συγκεντρώσει όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες, να εκπονήσουμε την έκθεσή μας. Η ιδέα τώρα εκπόνησης της έκθεσης αυτής έχει να κάνει πρώτον με το ότι θέλουμε συμμετοχή των εταίρων μας. Δεν θέλουμε εμείς να αφήσουμε απ' έξω κανέναν, ούτε να κάνουμε κηρύγματα σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να δούμε τα θέματα αυτά από πλευράς εσωτερικής αγοράς, πρώτα απ' όλα για να παρουσιάσουμε ποια είναι η παρούσα κατάσταση και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε συστάσεις. Τώρα, θέλουμε βέβαια να έχει νόημα η συμμετοχή των εταίρων μας. Διότι έχουμε βέβαια εμπειρογνώμονες και στις, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην αντιπροσωπεία μας για τις σχέσεις μας με άλλες χώρες. Αλλά όσοι δεν συμμετέχουν σε αυτά τα θέματα σε καθημερινή βάση μπορεί να έχουν μια άλλη οπτική γωνία και να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις τους με την εσωτερική αγορά. Θέλουμε να επικεντρωθούμε σε θέματα εσωτερικής αγοράς. Βλέπετε, μέχρι τώρα είχα συζητήσεις, διαβουλεύσεις με πρέσβεις και από την Ελβετία και από την Ορβηγία. Έχω μιλήσει και με εθνικούς βουλευτές, με την Κομισιόν και όταν φτάνουμε στα έγγραφα εργασίας μας λένε δεν είναι καλά ισορροπημένα, δεν δείχνουν ε, την ακριβή φύση των σχέσεών μας μαζί σας κλπ. κλπ. Λοιπόν τώρα θέλουμε να επικεντρωθούμε στην εσωτερική αγορά. Δεν μιλάμε για ολόκληρη τη δομή των σχέσεών μας, δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες για το πώς, πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις μας αυτές, αλλά προσπαθούμε με την έκθεση αυτή να επικεντρωθούμε όπως σας είπα στην εσωτερική αγορά, ε, βέβαια περνώντας και λιγάκι από τις γενικότερες σχέσεις μεταξύ μας. Θέλουμε μια συνεκτική έκθεση. Γιατί ξέρετε ότι δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, πολύ σέλιδη. Θα επικεντρωθούμε κυρίως σε συστάσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μερικές συστάσεις. Αλλά, όπως είπα πριν και το επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε να έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε με τους εταίρους μας όχι μόνο για το status quo, αλλά και για τα σημαντικά και δύσκολα θέματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Επιτροπή μας. Προστασία των καταναλωτών, ε, πακέτα κλπ. Και να, έχουμε εδώ τους πρέσβεις. Και αν δεν, απα... αν δεν απατώμε, έχουμε εδώ και από περιφερικά κοινοβούλια. Έτσι δεν είναι. Έτσι θα έχουμε και με εθνικούς βουλευτές ε, συζήτηση και από τις χώρες, δηλαδή ΕΟΧ, τους βουλευτές από τις χώρες ΕΟΧ. Η λέξη δυναμικό, δυναμισμός μπορεί να έχει και αρνητική χρειά από ό,τι κατάλαβα από συζητήσεις που είχα μέχρι τώρα μαζί σας. Εμείς λέμε θέλουμε να είναι όλοι, να έχουν δυναμική, αλλά κατάλαβα ότι ορισμένοι θεωρούν αρνητικό αυτόν τον όρο, γιατί σημαίνει ότι μειώνουμε την κυριαρχία των άλλων. Συνεπώς, η φύση των σχέσεών μας είναι δύσκολη και αυτό απορρέει από το γεγονός ότι οι Ελβετοί θέλουν να προστατεύουν την κυριαρχία τους, το οποίο σεβόμαστε απόλυτα βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ένα status quo και θέλουμε να μας πείτε, επιδέχεται βελτίωση ή όχι. Πρώτα απ' όλα θα μας παρουσιάσετε κάπως τη δομή, όπως ε, και ο καθηγητής και η καθηγήτρια Τόμπλερ ε, είπε θα ακούσουμε λοιπόν, ίσως πιο περιληπτικά, να σκεγγραφείτε την κατάσταση και μετά θέλουμε προτάσεις, συστάσεις. Για την τυποποίηση, για παράδειγμα, της διαδικασίας κοινοποίηση, για θέματα που έχουν να κάνουν με την έγκαιρη διαβίβαση εγγράφων. Να ακούσουμε και από τα κράτη-μέλη αλλά και από τις χώρες ΕΟΧ για τη Λισαβόνα που φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στα εθνικά κοινοβούλια. Τι πιστεύετε. Και μετά όταν πρόκειται για την αγορά επίσης. Υπάρχουν σχέσεις καλές, αλλά επιδέχονται πάντα βελτίωση, ακόμα και αν είναι πολύ καλές. Οι σχέσεις μας με την Ελβετία είναι βέβαια πιο περίπλοκες, πιο δύσκολες. Μπορούμε να συζητήσουμε κάποια θέματα από αυτού εδώ. Γιατί πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να κοιτάμε καλά το σύστημα και να αναρωτηθούμε. Μπορούμε να το βελτιώσουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε οι εταίροι μας να συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων, στη σκιαγράφηση των αποφάσεων. Να, κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν, μπορεί να μην είναι υπερβολικά φιλόδοξα. Και μετά υπάρχουν και πιο φιλόδοξα ζητήματα. Η υπογραφή συμφωνίας για τις υπηρεσίες ή συμφωνία πλαίσιο. Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε σε αυτήν. Η ακρόαση αυτή λοιπόν, αυτό το λόγο ύπαρξης έχει, να εντοπίζονται τα προβλήματα στο σύστημα, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα γιατί εγώ είμαι ειδικό κυρίω σε συνταγματικά ζητήματα και για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρω αυτά που λέτε για τα προηγούμενα που έχουμε, την απόφαση για το κασίς ε, της Διζών κλπ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγή που έκανες και ελπίζω ότι όλοι θα έχετε συνειδητοποιήσει ε, πόσο φιλόδοξο είναι το έγγραφο εργασίας ε, του Ραφάλ, γιατί έχετε συνεργαστεί ήδη μαζί του. Τώρα, κάποια τεχνικά, τεχνικά σημεία. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ε, αυτές τις ε, ε, κάμερες οι οποίες ανάβουν μόλις ανάβει και το μικρόφωνο σας. Γι' αυτό λοιπόν να είσαστε καλά τοποθετημένοι απέναντι στην κάμερα γιατί διαφορετικά θα βγάζει τον διπλανό σας και όχι εσάς. Επίσης να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά αναπαρέμβαση. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συνηθίσει να μιλάμε υπό την απειλή του ρολογιού και επομένως να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά. Ε, υπάρχουν ρολόγια στην αίθουσα και νομίζω ότι υπάρχει και ένα μπροστά σα που μετράει το χρόνο. Τώρα, θα έχουμε τέσσερις ε, παρουσιάσεις όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και ατόμων. Μετά θα δώσω, στο πάνελ, ε, θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μετά θα έχουμε με... και ενδεχομένως απάντηση από τους εμπειρογνώμονες. Μετά θα κάνουμε ε, ένα δεύτερο τμήμα που θα αφορά τις δημόσιες προμήθειες και μετά μια συζήτηση σε πάνελ ε, στο οποίο θα συμμετάσχει και η ε, κυρία Τόμπλερ καθώς επίσης και εκπρόσωπος του Λίχτενστάιν και οι εμπειρογνώμονες μας ελπίζω να συμμετάσχουν και στο πάνελ αυτό. Στη διάρκεια αυτού του τρίτου κομματιού, του τρίτου τμήματος, θα ασχοληθούμε και με πολιτικής φύσεως ζητήματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Έχουμε μαζί μας την κυρία Τρίνα Ράτμαν, η οποία είναι ε, υπεύθυνη, επικεφαλής μάλλον, της υπηρεσίας νορβηγικών επιχειρήσεων εις της ε, Βρυξέλλες, της ε, Ομοσπονδίας της Νορβηγίας. Επίσης πρέπει να καλωσορίσω και κάποια μέλη του Νορβηγικού Κοινοβουλίου τα οποία βρίσκονται εδώ μερικές ε, μέρες και παρακολουθούν και τις εργασίες μας. Έχουμε μαζί μας επίσης ε, την δόκτωρα Κριστίν ε, Καντούς από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Έχουμε τον κύριο Περ Νεστάντε ο οποίος είναι ιδιαίτερος γνωστός στην Επιτροπή μας γιατί ήταν πριν ε, μέλος ε, επιφανές της γραμματείας της Επιτροπής μας και ο οποίος τώρα εργάζεται για το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της χώρας του. Θα μας μιλήσει για την εφαρμογή της δέσμης ε, που αφορά τα αγαθά στις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ. Τέλος έχουμε τον κύριο Κλοντ Βίλντ, ο οποίος ε, είναι επικεφαλής της Ελβετικής Αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναφερθεί στην ε, αρχή του Κασίς του Ντιζόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας όσον αφορά την εφαρμογή της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες. Η Συνομοσπονδία των Νορβηγικών Επιχειρήσεων χαίρεται για την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αξιολογήσει την εφαρμογή της ε, οδηγίας για ε, την εσωτερική αγορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομική ανάπτυξη. Εδώ και 15 χρόνια με τη συμφωνία αυτή συμμετέχει η Νορβηγία στην εσωτερική αγορά και η συμφωνία αυτή έχει σχεδιαστεί πολύ καλά και μπορεί να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις, τις συνεχείς εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Νορβηγία βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο όσον αφορά το βαθμολόγιο για την εφαρμογή του δικαίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν λίγες ε, περιπτώσεις προσφυγής επί παραβάση εναντίον της Νορβηγίας. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο όμως βαθμολόγιο δείχνει ότι ο αριθμός των προσφυγών επί παραβάση έχει αυξηθεί κατά 32% σε σχέση με το προηγούμενο βαθμολόγιο και αυτό είναι κρίμα. Εμείς όμως είμαστε δεσμευμένοι υπέρ της ε, ελευθερίας με ελάχιστες απαιτήσεις από πλευρά των ε, οδηγιών και των κανονισμών. Η ελάχιστη εφαρμογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατερότητες των διαφόρων χωρών, γιατί αλλιώς υπάρχει υπερβολικό βάρος ε, σε βάρος των επιχειρήσεων. Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες Ξεκίνησε βέβαια μια τεράστια συζήτηση στην ε, Νορβηγία προκειμένου να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία ε, οι σχετικές διατάξεις. Εγκρίναμε ένα πλαίσιο στις 19 Ιανουαρίου του 2009. Η διαδικασία ελέγχου πάντως στην Νορβηγία δείχνει ότι υπάρχουν λίγες αλλαγές. Τέσσερις αλλαγές έχουν γίνει σε ειδικούς τομείς νομοθεσίας και υπάρχουμε μόνο ένα πρόγραμμα για άδειες που έχει αρθεί. Η Νορβηγία επίσης συμμετέχει και στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες ζητάει ότι οι απαιτήσει διατάξεις που έχουν ε, αρθεί να ε, υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε 73 authorization schemes τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση. Είναι υποχρεώσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Πρόκειται για το ειδικό επίπεδο, το εθνικό, το περιφερειακό, το τοπικό και αν συγκρίνουμε με τα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχει μεγαλύτερη συνδυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την οδηγία και τις απαιτήσει της. Η εφαρμογή λοιπόν έγινε έγκαιρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διοικητική ενσωμάτωση της οδηγίας έχει προχωρήσει επαρκώς. Όσον αφορά το ενιαίο σημείο επαφής, αυτό το φτιάξαμε με την δικτυακή μας πύλη Altin που συνδέεται με την δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Yugo. Έτσι έχουμε πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες απαιτήσει. Όμως η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, γιατί στο δικτυακό χώρο λέει ότι υπάρχει ένα ενιαίο σημείο επαφή όπου μπορούν να έχουν πληροφορίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να συλλέγουν ε, ενημέρωση, να μαθαίνουν τι αποφάσει υπάρχουν σε διάφορα διοικητικά επίπεδα. Όμως προ το παρόν δεν ανταποκρίνεται στον αρχικό στόχο γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι στα αγγλικά και δεν είναι πάρα πολύ εύκολη η πλοήγηση ώστε να μπορέσουν να έχουν τις απαντήσεις που θέλουν ε, οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, κάποιες αιτήσει υπάρχουν μόνο στα αγγλικά, κάποια έντυπα. Έτσι λοιπόν σήμερα το σημείο επαφής διευκολύνει πολύ λίγο την πρόσβαση στην αγορά της Νορβηγίας. Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες είναι ζωτικής σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν βέβαια προσπάθειες που συνεχίζονται ώστε το αυτό σημείο επαφής να γίνει αυτό που πρέπει σύμφωνα με την οδηγία. Η δεύτερη γενιά της δικτυακής πύλης Altin ακριβώς θα ξεκινήσει το 2011. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε ε, μεγαλύτερη επιτυχία. Πάντως θα πρέπει να υπάρχει ρητά κάτι που να βοηθάει την επίτευξη των στόχων, οι οποίοι εξάλλου δεν είναι αρκετά φιλόδοξοι πιστεύουμε. Οι υπηρεσίες, η ε, οδηγία για τις υπηρεσίες προσπαθεί να προχωρήσει χωρίς όμως να έχει γεωγραφικούς περιορισμούς. αν υπάρχει άρνηση μιας άδειας, αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται. Σύμφωνα με τις νορβηγικές διατάξεις, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με το άρθρο 13 πάντως της οδηγίας, ένας πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να παίρνει αυτόματα την άδεια εφόσον η προθεσμία έχει ξεπεραστεί. Αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 11 της ε, νορβηγικής πράξης όμως συνοδεύεται από το ότι unless otherwise stated by law or regulation, εκτός δηλαδή αν υπάρχει κάτι άλλο προβλέπεται από τον νόμο ή από κάποια, κάποιο κανονισμό. Το αποτέλεσμα είναι ότι δύο πράξεις οι οποίες έχουν ε, τροποποιηθεί για να ανταποκρίνονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες, δεν ε, ακολουθούν την πρακτική αυτή. Η οδηγία για τις υπηρεσίες λέει ότι το δικαίωμα για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά ε, ζητάει από τις κυβερνήσεις να φροντίσουν να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά, στην αγορά τους. Από την πράξη την ίδια. Όμως οι κυβερνήσεις ε, δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο ότι έχουν την υποχρέωση να το φροντίσουν αυτό, οι ίδιες οι κυβερνήσεις δηλαδή. Υπάρχουν απαιτήσει που οι κυβερνήσεις ε, τελικά δεν ακολουθούν. Η οδηγία για τις υπηρεσίε επίσης περιλαμβάνει πολλές διατάξει όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων. Υπάρχουν διατάξει που έχουν να κάνουν για την αμοιβαία αρρωγή, για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης όσον αφορά το νορβηγικό δίκαιο. όμω, η ε, ανταλλαγή αξιωματούχων δεν περιλαμβάνεται. Εμείς πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα ανταλλαγών θα βοηθούσε πάρα πολύ γιατί θα διευκόλυνε την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών και θα δημιουργούσε έτσι δίκτυα και ένα πιο ευρύ ε, δίκτυο επαφών. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αμοιβαία συστήματα. Αυτό θα βοηθήσει επίσης να γνωρίζει κανείς καλύτερα και τη συμφωνία με τον ΕΟΧ. Η Νορβηγία πιστεύει ότι υπάρχουν οικονομικοί, τεχνολογικοί και οι ανθρώπινοι πόροι για να τα καταφέρουμε καλύτερα όσον αφορά την ενσωμάτωση της οδηγία στην εθνική νομοθεσία. Πιστεύουμε όμως ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν δεσμευτεί επαρκώ. Εμείς είμαστε φιλόδοξοι, αλλά πιστεύουμε ότι το σημείο ενιαίας επαφής ε, δεν, δεν το έχουμε προσέξει όσο θα έπρεπε. Τα προβλήματα τα οποία εντοπίσαμε μέχρι τώρα συνοδεύονται και από τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, όπως είναι το πακέτο αγαθών. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό για βελτίωση εδώ. Εμεί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικέ κυβερνήσει θα πρέπει να κάνουν περισσότερε προσπάθειε για να ενημερώνουν τι επιχειρήσει, ιδιαίτερα τι μικρομεσαίε, για τα πλεονεκτήματα και τι ευκαιρίε που προσφέρει η οδηγία για τι υπηρεσίε ε, εφόσον εφαρμόζεται σωστά. Μια ιδιαιτερότητα για την ε, Νορβηγία υπάρχει και έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κοινοβούλιο μας δεν ενημερώνεται συγχρόνως με όλα τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς υποστηρίζουμε το σχόλιο του κύριου Τρασκόφσκη πριν από λίγο ότι το Νορβηγικό Κοινοβούλιο και όλα τα κοινοβούλια όχι πρέπει να ενημερώνονται συγχρόνως όπως και τα κράτη-μέλη, όπως και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Έτσι θα προχωρήσει πιο γρήγορα η ενσωμάτωση τη κοινοτικής ε, νομοθεσίας στην ε, εθνική μας, στην Ορβηγία. Τέλος θέλουμε να επαναλάβουμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που δίνεται τη σημασία αυτή στην Συμφωνία ΕΟΧ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Εσωτερική Αγορά. Αν δεν γνωρίζουμε καλά την συμφωνία ε, με τις χώρες ΕΟΧ, καταλαβαίνετε ότι έτσι δυσκολεύονται οι συναλλαγέ, δυσκολεύεται η πρόσβαση στην αγορά μα. Ο κόσμο λοιπόν πρέπει να γνωρίζει, οι επιχειρήσει και οι πολίτε πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία με τι χώρε ΕΟΧ. Ε, νομίζω ότι η ενίσχυση της ενημέρωσης όσον αφορά τη Συμφωνία ΕΟΧ από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί για να μην υπάρχουν πια εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ράτμαν για όλα αυτά τα, τον εξαντλητικό τρόπο μάλλον τον οποίο ε, αναφερθήκατε στο θέμα που μας ε, απασχολεί. Σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήματα τα οποία θα δούμε απέναντι. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στις 27 Απριλίου θα έχουμε μαζί με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων κοινή συνεδρίαση όσον αφορά ακριβώς την εφαρμογή της ε, ε, οδηγίας ε, για την κυκλοφορία των αγαθών. Και πραγματικά σας καλώ να είστε παρούσα στην ανταλλαγή απόψεων που θα λάβει η χώρα τότε και επίσης θα έχουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος ε, θα πάρει τον ε, λόγο γιατί βεβαίως και υπό το φως της νέας ε, συνθήκης της Λισαβόνας τα πράγματα έχουν αλλάξει και χρειάζεται και η συνένεση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος όλα αυτά που συζητούμε για την εσωτερική αγορά να μην κοινοποιούνται και στις χώρες ΕΟΧ και ΕΖΕΣ. Ελεύθερη κυκλοφορία ε, προσώπων και δίνω το λόγο στην κυρία Κριστίνη Καντού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Η Συμφωνία για την Ελεύθερη Κυκλοφορία ε, των Ατόμων ε, είναι μια συμφωνία του 99 που τέθηκε σε ισχύ το 2002. Επομένως ε, ισχύει εδώ και 8 χρόνια και στόχο έχει την ελεύθερη κυκλοφορία των, ε, των ε, ατόμων με τρόπο βαθμιαίο ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία. Μία από τις βασικές αρχές της συμφωνίας αυτής που ήδη έχει αναφερθεί είναι ότι δεν ενστερνίζεται ε, το κοινοτικό κεκτημένο. Δηλαδή δεν μεταφράζονται απολύτως οι αρχές της εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για μία συμφωνία η οποία θα δημιουργήσει δίκαιο παρόμοιο ε, με ε, αυτό που δημιουργείται όσον αφορά την νομοθεσία και την νομολογία η οποία δημιουργείται και απορρέει ακριβώς από την υπογραφή της συμφωνίας. Βεβαίως το σύστημα άρχισε να εφαρμόζεται ε, με δυνατότητα βαθμιαίας προσαρμογής. Η προσαρμογή όμως η οποία προβλέπετε δεν είναι αυτόματη. Βεβαίως υφίσταται μέσω ενός μηχανισμού που φέρει το όνομα μικτής, ε, ε, Μικτή Επιτροπή. Στη Μικτή αυτή Επιτροπή λοιπόν τα συμβαλόμενα μέρη σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορούν να προσαρμόσουν τα παραρτήματα κυρίως υπαριθμών 2 και 3 που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και την αναγνώριση των διπλωμάτων. Είναι γεγονός ότι οι αρμοδιότητες είναι περιορισμένες. Εάν θέλουμε να προσαρμόσουμε τις ε, διατάξεις ε, του σώματος του κειμένου και του παραρτήματος 1 θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί το σύνολο του κειμένου ε, πράγμα που σημαίνει διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και επιμέρους με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η διάρθρωση, η ίδια η φύση της ε, συμφωνίας ε, προκαλεί ε, τα, εμπόδια και τις δυσκολίες τα οποία έχουμε αναφέρει στο έγγραφο το οποίο έχουμε προετοιμάσει. βεβαίως λοιπόν εν συμπεράσματι μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρξει προσαρμογή αλλά είναι περιορισμένη. Η συμφωνία αυτή λοιπόν θα βασιστεί σε διατάξεις ε, οι οποίες ήδη υφίστανται στα πλαίσια της συνθήκης και που όμως έχουν προσαρμοστεί στις ε, διμερείς ε, σχέσεις της Ελβετίας βασιζόμενη βεβαίως σε αυτή την αρχή της ισοτιμίας της νομοθεσίας. Η συμφωνία αυτή αποσκοπεί στο να δοθεί αφενός άδεια παραμονής και εργασίας για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή είναι η καρδιά, αν θέλετε, ο πυρήνας ε, της ε, συμφωνίας και βεβαίως το τμήμα των υπηρεσιών, το οποίο όμως αναπτύσσεται πολύ λιγότερο στα πλαίσια αυτής της διμερούς συμφωνίας, γιατί στοχεύουμε στην απελευθέρωση ε, των δραστηριοτήτων για μια πολύ μικρή χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Τώρα, το τμήμα των ε, ε, υπηρεσιών είναι κάτι διαφορετικό και καλύπτεται μονάχα εν μέρη από αυτήν την, ε, αυτή την διμερή συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, προσώπων. Επομένως, κατά αυτήν την έννοια έχουμε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον πάροχο της υπηρεσίας. Εν προκειμένου, ο πάροχος μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του στο έδαφος της μίας ή της άλλης χώρας Εφαρμόζονται λοιπόν οι διατάξεις έτσι όπως εφαρμόζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είναι ενδιαφέρον να δει κανείς ε, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών είναι ότι επιτρέπει άσκηση δραστηριότητας όχι μονάχα στα, στα φυσικά πρόσωπα αλλά και στα ηθικά πρόσωπα πράγμα που δεν ε, συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε και μάλιστα απόφαση του δικαστηρίου Φεβρουαρίου του 2010 η οποία αναφέρει ότι ε, η κατάσταση διαφέρει αν μιλάμε για, ηθικά, για φυσικά ή για ε, ηθικά πρόσωπα και εν προκειμένου επρόκειτο για αγοραπολισία ακινήτου ή στην Αυστρία. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα ε, για αυτά τα μη φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ε, ε, συμπεριλαμβάνονται σε άλλη περίπτωση. Όσον αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, βεβαίως τα κεντρικά θέματα εδώ είναι η δραστηριότητα των ε, μετατοπισμένων εργαζόμενων. Ε, υπάρχει λοιπόν μια διάταξη η οποία δίνει τη δυνατότητα στα συμβαλόμενα μέρη να αναλάβουν ε, νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις προβλέψεις των, για τα δικαιώματα των εργαζομένων και επομένως στο παράρτημα 1 υπάρχει μια διάταξη που επιτρέπει στα εμπλεκόμενα μέρη να ε, αναλάβουν ε, ε, να λάβουν αποφάσεις βάσει της ε, οδηγίας του 96 αποφεύγοντας βεβαίως το κοινωνικό ή το μισθολογικό dumping. Πρέπει να πούμε ότι μετά τη συμφωνία του 96 υπήρξαν και κάποια συνοδευτικά μέτρα. Η διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων, ο καθορισμός ε, του ύψους των μισθολογικών ε, απαιτήσεων αναέτος και βεβαίως ένα τρίτο σκέλος όσον αφορά... Euh, ε, όσον αφορά τους αποσπασμένους ε, υπαλλήλους, σχετικά δηλαδή, εργαζόμενους, σχετικά δηλαδή με το χρόνο εργασίας τους, την ε, αμοιβή τους κτλ. Βεβαίως, ε, πριν από την αρχή της απόσπασης, ε, ο εργοδότης οφείλει να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απόσπασης, τον αριθμό των υπαλλήλων κτλ. Εδώ υπήρξε επίκριση ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανόνα των λεγόμενο κανόνα των 8 ημερών. Δηλαδή, ο εργοδότης έχει την ε, ε, δυνατότητα να αποφασίσει ότι οκτώ μέρες μετά την ανακοίνωση της απόσπασης και αυτού του είδους παροχής υπηρεσίας μπορεί να αρχίσει η ίδια η παροχή υπηρεσίας. Υπάρχει λοιπόν ένας κανόνας ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ε, περιορισμός της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Όμως, όμως, θα πρέπει κανείς να επαληθεύσει εάν ο στόχος, ο επιδιωκόμενος στόχος, ο στόχος λοιπόν που επιδιώκεται από το μέτρο αυτό είναι αρκετά δικαιολογημένος. Ε, εάν δηλαδή ο κίνδυνος κοινωνικού ή ε, μισθολογικού ντάμπινγκ επιτρέπει την χρήση αυτού του μέτρου και δεύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει ε, να συζητηθεί εάν απαντήσουμε ε, θετικά στο πρώτο ερώτημα, στην πρώτη υπόθεση, είναι να δούμε εάν υπάρχει αναλογικότητα στο μέτρο αυτό. Το ζήτημα είναι ανοιχτό, δεν έχει υπάρξει απόφαση ε, νομική, όμως ε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι εάν πρόκειται για περιορισμό ε, θεωρούμε ότι σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία ήδη περιέχονται στην ονομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτός ο περιορισμός είναι θεμητός και επίσης όσον αφορά τον περιορισμό αυτών των οκτώ ημερών τι να σας πω, ε, πρόκειται το θέμα των αποσπασμένων εργαζόμενων ε, είναι ευαίσθητο και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ανακοίνωση της Επιτροπής του 2007 που αναφέρεται στα προσκόμματα ε, τα οποία παρουσιάζονται στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και είναι γεγονός ότι ακόμα και οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρόβλημα με αυτή την ρήτρα αναγγελίας της απόσπασης. Πράγμα σημαίνει ότι γενικότερα ε, αυτό το ζήτημα είναι προβληματικό. Πάντως το θέμα δεν έχει απαντηθεί οριστικά και νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε στο πάνελ το θέμα αυτό αργότερα, αλλά στην ουσία απλώς αυτός ο κανόνας των οκτώ ημερών ε, μικραίνει όλο και περισσότερο. Επίσης, η χρηματική ε, ρήτρα, η οποία, αυτή η χρηματική εγγύηση βάσει του κανονισμού της Βασιλείας, αυτή, η, αυτός ο κανόνας έχει ε, εφαρμοστεί hm, αρχικά στην Ελβετία, ενώ το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους κατηργήθη, στην ουσία μετά από αποφάσεις του δικαστηρίου. Πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει ερμηνευθεί διαφορετικά από τα ελβετικά δικαστήρια. Πάντως πρέπει να πούμε ότι οι ε, διατάξεις σχετικά με τους αποδέκτες ε, ε, υπηρεσίας είναι διαφορετικές είναι διαφορετικές στην ε, Ελβετία από ότι ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να επανέλθουμε πάνω σε αυτό. Ορισμένα συμπεράσματα. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της συμφωνίας οπωσδήποτε έχει πιο περιορισμένο εύρος από αυτό που έχει στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποτελεί πλήρη απελευθέρωση της κυκλοφορίας των ατόμων και οι δυσκολίες οι οποίες διεφάνησαν κατά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας είναι ε, συγκεκριμένες και μεμονωμένες μπορώ να πω ότι οι μείζονες δυσκολίες οι οποίες παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή ε, της ε, συμφωνίας στην, οποία, ε, στην ουσία είναι εγγενείς προς την, προς την φύση της συμφωνίας και προς τους μηχανισμούς εφαρμογής όμως δεν αφορούν την ιδιαίτερη μορφή εφαρμογής. Αφορούν στην ουσία δηλαδή το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ την uh, κυρία Καντού για την παρουσίασή της. Και ευχαριστούμε που αναφέρατε κάποια φλέγοντα θέματα όπως αυτό της απόσπασης των εργαζομένων που είναι και σημαντικό και για, την, uh, τον ΕΟΧ και για την Ελβετία και για την δική μας ε, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και σημαντικό σημείο στην ε, μοιραστή διάταξη για, την, για τον Επίτροπο Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Άντορ. Um, Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ Εγώ εργάζομαι στο Υπουργείο Εμπορίου και Ανάπτυξης ε, και ασχολούμαι με θέματα ε, εσωτερικής αγοράς, εμπορίου, μετάθεση των απόσπαση των ε, εργαζομένων; Ευχαριστώ για την ίδια πρωτοβουλία και για την έκθεση και για και τον εισηγητή. Και θα ήθελα όντω να μπορέσουμε να συζητήσουμε σήμερα το θέμα τη ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, που είναι μία από τι βασικέ ελευθερίε τη εσωτερική αγορά. Κάποια βασικά σημεία θα ήθελα να σα αναφέρω σήμερα. Η εσωτερική αγορά είναι πολύ σημαντική για την ε, Νορβηγία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακράν ε, ο μεγαλύτερο εταίρος μα εμπορικός μας 70% των εισαγωγών μα και 80% των εξαγωγών μα προέρχονται από εδώ. Και πιστεύουμε ότι το πακέτο αυτό θα ε, βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα των αγορών η δημιουργία των ενιαίων σημείων επαφής είναι πολύ σημαντικά επίσης ως προς την επίτευξη του σκοπού αυτού και Πρέπει να προχωρήσουμε με την εφαρμογή του πακέτου. Για να σεβαστούμε όμως ε, και τι ε, εθνικέ νομοθεσίες θα χρειαστεί χρόνος. Αλλά έχουμε στόχο την πλήρη ε, εφαρμογή άπαξ, διαπαντός. Οπότε πρέπει να γίνουν και οι αναγκαίες αλλαγές για να γίνει αυτό. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και στα πλαίσια της Κομισιόν ως προς αυτό και βεβαίω στην όλη συζήτηση παίρνουν ε, ε, μέρο και οι χώρε ΟΧ ε, και έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των προτάσεων που υποβάλλονται. Η πρόταση αυτή για το πακέτο για τα αγαθά μπήκε σε δημόσια διαβούλευση στην Νορβηγία ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση και να εξασφαλίσουμε ότι τα σημαντικά θέματα και τα συμφέροντα θα εκπροσωπούνταν πλήρω και θα τα λαμβάναμε υπόψη. Υπήρξε γενική ε, υποστήριξη και το βασικό ήταν ε, αυτό στην ε, διάσκεψη που έγινε. Δώσαμε εμείς την άποψη στο Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2007. Το 2007 έγινε ένα, μια διυπουργική... Ε, συγγνώμη, η, διερμηνείς δυσκολεύονται να σας παρακολουθήσουν. Μήπως μπορείτε να τα πείτε λίγο πιο αργά. Συγγνώμη. Και αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να μιλάτε. Um, το 2007 έγινε μια, ε, ένα, μια ομάδα εργασία στην Υπουργική, ad hoc, για να, δημιουργηθεί, για να διευκολυνθεί η ε, ανταλλαγή πληροφοριών και η κοινή κατανόηση του πακέτου σε όλα τα επίπεδα τη ε, διακυβέρνηση. Μετά από την επίσημη έγκριση αυτού του πακέτου, ε, το Υπουργείο ξεκίνησε να κάνει τι απαραίτητε αλλαγέ ε, στην ε, ε, νορβηγική ε, νομοθεσία. Αυτό θα γίνει μέσω δύο νομικών πράξεων, μία για κάθε κανονισμό. Ε, μια ευρεία δημόσια διαβούλευση για τι δύο αυτέ πράξει έχει προετοιμαστεί από, το, από, το από την ομάδα εργασία του Υπουργείου του Νορβηγικού. Το έγγραφο αυτό κυκλοφόρησε 8 Φεβρουαρίου φέτο με μια περίοδο διαβούλευση τριών μηνών. Μετά την, ε, το, την ολοκλήρωση τη διαβούλευση, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα και θα προετοιμάσουμε μια λευκή βίβλο για το ε, Νορβηγικό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι οι τελικές πράξει θα μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ στι αρχές του 2011. Όπως είπα, έχουμε στόχο στην πλήρη ε, ε, εφαρμογή και, του, και των νεοδιοικητικών συστημάτων και των δύο νομικών πράξεων. Παράλληλα με την εθνική ε, εφαρμογή και την όλη διαδικασία, οι χώρε ΟΧΕΖΕ εργάζονται ω προ την εφαρμογή, ω προ την ενσωμάτωση των δύο κανονισμών στην, στην Συμφωνία ΕΟΧ. Όπω είπα, πιστεύουμε ότι οι νέοι κανόνε θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των αγορών και στα πιο ασφαλή προϊόντα. Φυσικά, οι νέοι κανόνε έχουν ω στόχο να ενισχύσουν την εποπτεία τη αγορά. Στην Ορβηγία προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα ένα, μια ομάδα εποπτείας υπουργική, εποπτείας της αγοράς, που θα, της οποίας θα προεδρεύει το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η ομάδα θα εξασφαλίσει τον συντονισμό και θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσει γίνονται σεβαστές σε ό,τι αφορά τον κανονισμό. Δύο υπάρχοντα ε, δίκτυα για, την, ε, για τις αρχές εποπτείας θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να, ε, είναι, να λογοδοτούν στην συντονιστική ομάδα. Επίση, θα δημιουργήσουμε τα προγράμματα που προβλέπονται στον κανονισμό και στην παρούσα διαβούλευση ζητούμε ε, συμβολή, ε, είτε είναι οριζόντια είτε τομεακή, ή συνδυασμό και των δύο. Ε, καλωσορίζουμε μια πιο συγκεκριμένη στοχοθέτηση στην αποκτήρια τη αγορά στην εσωτερική αγορά και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι κάθε ε, χώρα πρέπει να αναλάβει το δικό τη μερίδιο ευθύνη έτσι ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Θεωρώ ότι η ΙΜΚΟ μπορεί να παίξει ένα ρόλο ώστε να ενθαρρύνει τα κρατημέλη να αναλάβουν τη δική του ευθύνη προ αυτό. Χαιρόμαστε που βλέπουμε την ενίσχυση τη ευρωπαϊκή πιστοποίηση ω αποτέλεσμα του πακέτου για τα αγαθά και επίση ότι η τυποποίηση είναι ένα ε, χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία τη εσωτερική αγορά. Το Κοινοβούλιο, ή η Κομισιόν, συγγνώμη, ε, εμπλέκεται στην όλη η κομισιον συγγνωμη μπλέκεται στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Συστήματο Τυποποίηση. Εμεί υποστηρίζουμε το στόχο αυτό και θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και στα πλαίσια των συζητήσεων που γίνεται για το πακέτο ε, τυποποίηση που προετοιμάζεται από την Κομισιόν. Ω μη μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό αποτελεί καμιά φορά πρόκληση και θα ήθελα να σα αναφέρω κάποια παραδείγματα που ανέφερε και η προηγούμενη καθηγήτρια και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Οι κανονισμοί είναι προτιμόμενο εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσουν τους, ε, ότι οι κανόνε θα, ε, θα τεθούν γρήγορα σε ισχύ. Βέβαια, ε, από την πλευρά τη ΟΧΕΖΕΣ, η διαφορά μεταξύ κανονισμών και, και οδηγιών είναι λιγότερο σημαντική. Εμεί χρειαζόμαστε να πρέπει να εφαρμόσουμε και τα δύο αυτά εργαλεία στο δικό μα εθνικό δίκτυο και είναι δύσκολο καμιά φορά να εξασφαλίσουμε ότι τίθενται σε εφαρμογή οι, οι κανονισμοί τον ίδιο, την ίδια ώρα. Τώρα, οι συζητήσει στο Συμβούλιο και στι ομάδε εργασία του και οι άτυποι, οι άτυποι τριμερεί διάλογοι είναι, δεν είναι ανοιχτοί σε μη μέλη, αλλά αυτό σημαίνει ότι μετά την επίσημη έγκριση των, του πακέτου για τα αγαθά ε, είχαμε, έπρεπε να εξετάσουμε τα τελικά κείμενα προσεκτικά ε, ώστε να ξέρουμε αν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στο, ε, στην εθνική μα νομοθεσία. Επίση, η ευαισθητοποίηση. Ξέρουμε ότι κάποιε νορβηγικέ επιχειρήσει αντιμετωπίζουν εμπορικά εμπόδια λόγω του ότι οι αρχέ στα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν ακριβώ την συμφωνία ΕΟΧ και, δεν, και ότι η Νορβηγία είναι μέρο τη ιστορική αγορά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και είναι, και, ο λόγο για τον οποίο το Solvit και άλλα εργαλεία μπορούν να μα βοηθήσουν ω προ αυτό. Επίση, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μεταξύ τη Κομισιόν και τη ε, Αρχή Εποπτεία τη ΕΦΤΑ, τη ΕΖΕΣ, για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων κανόνων. Τέλο, να σα θυμίσω ότι οι χώρε ΕΖΕΣ δεν είναι, μέρος, δεν είναι τμήμα τη Ελληνική Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχέ λοιπόν που είναι υπεύθυνε για τι αρχέ ε, για τον εξωτερικό έλεγχο ε, προβλέπεται να έχουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των αγαθών ώστε να μην μπαίνουν επικίνδυνα αγαθά στην εσωτερική αγορά. Τα αγαθά που δεν ε, μπαίνουν στην εσωτερική αγορά, ε, θα πρέπει να, στην εσωτερική αγορά τη Ένωση, θα πρέπει να απαγορεύεται να μπαίνουν και στι χώρε Εζέ. Η στενότερη λοιπόν συνεργασία και συντονισμό θα πρέπει, να, είναι, θα πρέπει να, ισχύ, να υπάρξει για να, αντιμετωπιστούν αυτέ οι προκλήσει. Να πω ότι η δουλειά για το πακέτο για τα προϊόντα έχει, γίνει μεγάλη, έχει αποτελέσει την ευκαιρία για να έχουμε καλύτερη ευαισθητοποίηση και ότι σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και αγαθών ε, στι εθνικέ κυβερνήσει και στου υπόλοιπου φορεί. Η Νορβηγία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την πλήρη θέση σε εφαρμογή των, ε, του πακέτου όσο δυνατόν πιο σύντομα. Ε, θα, αναλάβουμε τα απαραίτητα, θα αναλάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί επισήμω και στον εθνικό μας, ε, στην εθνική μα νομοθεσία, αλλά θα κάνουμε και τι απαραίτητε αλλαγέ που χρειάζονται για να λειτουργήσει το σύστημα. Εγώ προσβλέπω στην έκθεση του εισηγητού και βεβαίω αν υπάρχουν ερωτήσει ή αν θέλετε περισσότερε πληροφορίε, ευχαρίστω να σα απαντήσω. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι υπάρχουν ακόμα και πολλά φλέγοντα ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και τα οποία είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη των εργασιών μας όσον αφορά την επιστοποίηση όσον αφορά επίσης την εφαρμογή της δέσμης των αγαθών. Ο η συγητή μου ζήτησε συγγνώμη, ε, θα πρέπει να δώσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση ε, και θα επιστρέψει αμέσως. Ε, θα του πούμε τι συνέβη, θα του κάνουμε ένα briefing. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στον κύριο Κλοντ Βίλντ από την Ελβετική Αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας μιλήσει για την αυτόνομη εισαγωγή της αρχής του Κασίς Ντοντιζόν. Πρόσφατες εξελίξεις και ε, μελλοντικές προκλήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, στα πλαίσια τη παρούσα ακρόαση, σα ευχαριστώ που βάλατε στη μέρη σε διάταξη το θέμα τη μονομερού εισαγωγή τη αρχή Κασί Ντοντιζόν στην Ελβετία. Όντω, το θέμα αυτό επιτρέπει ε, να αποδειχθεί ότι η Ελβετία είναι ένας εταίρος ο οποίος θέλει να προωθήσει την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αποτελεί πηγή προβλημάτων και δυσκολιών στην εφαρμογή της προαναφερθήσης. Στις 12 Ιουνίου 2009 το Ελβετικό Κοινοβούλιο αποφάσισε ε, την πλήρη ε, μονομερή εφαρμογή της αρχής Κασίς Dijon αναθεωρώντας τον ομοσπονδιακό νόμο όσον αφορά τα τεχνικά προσκόμματα ε, προς το εμπόριο. Αυτή η αναθεώρηση δίνει την δυνατότητα στα περισσότερα προϊόντα τα οποία νομίμως τίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες ΕΖΕΣ δίνει τη δυνατότητα λέγω να κυκλοφορήσουν ελεύθερα και στην Ελβετία. Η προϋπόθεση Βεβαίω είναι να μην παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα όσον αφορά το ιδιαίτερο δημόσιο συμφέρον, κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Ε, επομένως, προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν ε, διμερείς ε, συμφωνίες ε, και δεν υπάρχουν εναρμονισμένες αρχές για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κυκλοφορούσουν ελεύθερα στην ελβετική αγορά. Αναφέρομαι κυρίως σε καλλιντικά υφάσματα ή διένδυσης και έπιπλα. Όσον αφορά τώρα τα τρόφιμα, η αναθεώρηση του νόμου προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς που επιτρέπει την μονομερή εφαρμογή της αρχής του Cassis de Dijon υπό την αίρεση μιας ειδικής άδειας από, το, από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας. Η άδεια αυτή ε, δίνεται για τα τρόφιμα τα οποία παράγονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ε, της ε, συνθήκης ΕΖΕΣ. Μονάχα λοιπόν πολύ μικρός αριθμός προϊόντων αποκλείονται, περίπου 20. Η, κύριε Πρόεδρε, η μονομερής εφαρμογή τη αρχής ε, του Cassis de από την Ελβετία αντιπροσωπεύει ένα νέο μέτρο το οποίο θέλει να άρει τι ε, τεχνικές ε, δυσκολίε και τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης επιτρέπει ε, στην Ελβετία να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πολιτική και επομένως να συμβάλλει στην μείωση των προϊόντων ε, κατανάλωσης. Η προσπάθεια μείωσης ε, των υψηλών τιμών πρόκειται, είναι, αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της ελβετικής κυβέρνησης και βεβαίως πέρα από αυτή την υπολογιζόμενη επίπτωση όσον αφορά την μείωση των τιμών μπορώ να σας εξηγήσω γιατί η Ελβετία αποφάσισε να εφαρμόσει μονομερώς αυτήν την αρχή του de Dijon. Όντως συνήθως το άνοιγμα της αγοράς μιας χώρας υπέρ ενός εταίρου γίνεται σε αμοιβαία βάση. Εδώ μπορώ να σας απαντήσω με δύο τρόπους. Πρώτον, αυτή η αναθεώρηση αφορά και συνεχίζει την παράδοση ανοίγματο της Ελβετίας ε, σε σχέση με τις εμπορικές της ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ιδιαίτερο μέτρο, η Ελβετία έλαβε επίσης υπόψη της ε, τις διαπραγματεύσεις ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των αγροτικών και προϊόντων και των προϊόντων διατροφής. Αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν προετοιμαστεί επί ε, πολλά έτη και συγκεκριμένα ξεκίνησαν από τον Νοέμβριο του 2008. Τροποποιώντας μονομερώς τον Ομοσπονδιακό Νόμο όσον αφορά τα τεχνικά προσκόμματα ε, προς το εμπόριο, η Ελβετία εκ των προτέρων ε, προδικάζει την ε, πλήρη και αμοιβαία απελευθέρωση των ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στον εναρμονισμένο και τον μη εναρμονισμένο τομέα των ε, γεωργικών και προϊόντων και προϊόντων διατροφής. Είναι αυτονόητο ότι βεβαίως η Ελβετία περιμένει και από τους Ευρωπαίους εταίρους την αμοιβαία αναγνώριση των προσπαθειών αυτών. Ε, και βεβαίως ε, αυτό ε, σημαίνει ότι με την εφαρμογή της συνθήκης η οποία τώρα βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση τα ευρωπαϊκά προϊόντα οπωσδήποτε θα κυκλοφορήσουν ελεύθερα στην ελβετική αγορά. Στα πλαίσια των προαναφερθισών διαπραγματεύσεων δεν έχουν ακόμα δοθεί από την ε, Κομισιόν στην Ελβετία η τα προσδοκόμενα εχέγγυα αμοιβαιότητα. Αυτό μας λυπεί ιδιαιτέρως, διότι για την Ελβετία κύριος στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η αμοιβαία δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές των δύο εταίρων, καθώς επίσης και η κατάργηση των περισσότερων ελέγχων στα σύνορα. Για την ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται σε μια ολοκλήρωση του μη εναρμονισμένου το τομέα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Εμείς θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλα τα προϊόντα της διατροφικής γεωργικής αλυσίδας και θα πρέπει να οδηγήσει σε πλήρη άρση και κατάργηση όλων των εμποδίων στο εμπόριο. Είτε πρόκειται για δασμολογική ε, για δασμολογικά είτε μη δασμολογικά ε, προβλήματα. Η ολοκλήρωση μια τέτοια συμφωνία θα επιτρέψει και την ολοκλήρωση τη απελευθέρωση του εμπορίου των γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων μεταξύ τη Ελβετία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό προ το αμοιβαίο συμφέρον των δύο πλευρών. Ολοκληρώνοντα, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω ότι και θέλω να, το, να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να δούμε την πολιτική σημασία της μονομερούς εφαρμογής της αρχής του Cassis de Dijon από την ε, Ελβετία και τις πολιτικές του προεκτάσεις. Όπως έλεγα και στην αρχή της παρέμβασής μου, αυτό το μονομερές μέτρο καταδεικνύει ότι η Ελβετία δεν αποτελεί πηγή προβλημάτων και προσκομμάτων στην ελεύθερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αντιθέτως, θέλει να ενισχύσει την ε, δράση και το πεδίο εφαρμογής της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ σαφή ε, εισαγωγή που μας κάνατε όσον αφορά την μονομερή εισαγωγή αυτού του πολύ ε, σημαντικού θέματος της αρχής ε, του Κασίς ε, Ντιζόν. Είμαι σίγουρη, σίγουρος συγγνώμη, ότι θα έχετε πολλές ερωτήσεις να υποβάλλετε. Έχουμε λίγα λεπτά πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο τμήμα Ενδεχομένως ο εισηγητής θα ήθελε να κάνει κάποια σχόλια και δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος να υποβάλει κάποια ερώτηση. Δεν έχουμε βέβαια πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και πρέπει να συνεχίσουμε με το δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Αλλά ενδεχομένως ο εισηγητής θα μπορούσε να κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι και εμείς χρησιμοποιούμε τη δυναμική στην προσέγγισή μας και όσον αφορά την υπόθεση του Κασίς της Τιζών θα μπει στην έκθεση. Είχαμε ένα έγγραφο εργασίας, τώρα ετοιμάζουμε μια έκθεση. Αυτή είναι η δυναμική στη διαδικασία. Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι για τα μέτρα στήριξης. Εμείς καταλαβαίνουμε γιατί μερικά από τα μέτρα στήριξης υπάρχουν κοινωνικό ντάμπινγκ και άλλα. Όμως, άσο, ξέρω, το θέμα είναι το θέμα της αναλογικότητας. Γιατί σύμφωνα με το CGA, το θέμα αυτό θα ήταν αποδεκτό εφόσον γίνεται σεβαστή η αναλογικότητα και αν αποδεικνύεται ότι το γενικό συμφέρον δεν καλύπτεται αρχικά. Οπότε αυτό είναι το κύριο θέμα που μας απασχολεί δεν είναι ότι πάντα κριτικάρουμε οποιοδήποτε μέτρο στήριξης. Όχι. Αυτό που ρωτάμε είναι, είναι αναλογικό. Και αυτή είναι η ερώτησή μου. Εσείς πώς το αξιολογείτε αυτό. Έπειτα, στην έκθεσή μας σημειώνουμε ότι δεν είναι μονόδρομος, ότι υπάρχουν προβλήματα που έχουν οι οικονομικοί μας εταίροι στην Ελβετία, αλλά βλέπετε ότι οι Ελβετοί έχουν προβλήματα, αλλά έχουμε και εμείς στις χώρες μας. Όταν, για παράδειγμα, συζητάμε θέματα όπως είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών, και εμείς τα έχουμε στις χώρες μας, στις χώρες μέλη για την παροχή υπηρεσιών. Δεν είναι κάτι καινούριο, όμως το δικό μας το σύστημα Πρώτα απ' όλα πάντα μπορούμε να βασιστούμε στους κανονισμούς του CGA και πάντα ε, εξετάζουμε και το θέμα της αναλλαγικότητας. Αυτή λοιπόν είναι η δυσκολία. Δεν είναι ότι εμείς λέμε Α, ό,τι κανόνες εσείς ε, βάζετε δεν ε, αιτιολογούνται. Όχι. Απλώς δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτή τη δοκιμή για να δούμε είναι αναλογικά ή δεν είναι. Ο Άντρες θέλει να πάρει το λόγο, ο θέλει να πάρει το και μετά ίσως και η Επιτροπή να απαντήσει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε. Οι παρουσιάσει ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Όντω, σε πολλά σε πολλά θέματα έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα που τα έχουμε συζητήσει και στα κράτη-μέλη. Και για τον ΕΟΧ και για την ε, Ελβετία. Έχω ένα ερώτημα για τον ε, κύριο Βίλντ, ο οποίο ε, μίλησε για μονομερέ άνοιγμα τη αγορά και με την ομολογία για το Cassis de Dijon αυτή η, αυτό, αυτή η μονόπλευρη προσέγγιση ισχύει δεν ισχύει για όλα τα κράτη. Δηλαδή η Ελβετία σήμερα έχει πρόσβαση στις αγορές πολλών κρατών μελών με τα, με τα προϊόντα της. Ε, και θα ήθελα και την, για την κυρία Καντής να ρωτήσω. Αναφέρε, αναφέρετε κάτι για την ε, προ... Ε, ανακοίνωση Είπατε ότι το πρόβλημα προέκυψε γιατί το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας ε, και οδήγησαν, αλλά και οι μηχανισμοί, οδήγησαν στο να μην υπάρχει διαφορετική ε, δυνατότητα, διαφορετικός δρόμος. Δεν υπάρχουν δηλαδή καμία άλλη, δεν υπάρχει κανένα, καμιά άλλη ενακτική. Right. Um, Καλώς. Ποιος θα ξεκινήσει. Ε, η καθηγήτρια Καντούς ίσως πρώτα. Ο κύριο Στρακόφσκι εσάς ρώτησε και τον κύριο Βιτς βέβαια και η καθηγήτρια Τέμπλερ θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Για τα μέτρα αυτά τα συνοδευτικά. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελβετία και στο κάτω-κάτω σε κάθε διμερή σχέση με μια χώρα όπου τίθεται θέμα παροχής υπηρεσιών. Το θέμα είναι, δικαιολογείται το μέτρο. Και το άλλο είναι η αναλογικότητα. Σε ένα σύστημα έτσι όπως αναπτύχθηκε από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εννοείται ότι υπάρχουν διάφορα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί και καλώς. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε εσείς είναι ότι στα πλαίσια της διμερούς συμφωνίας έχετε ένα σύστημα ρύθμισης των διαφορών, διευθέτησης των διαφορών, εποπτείας αν θέλετε εφαρμογής της συμφωνίας που γίνεται μέσω μιας μικτής επιτροπής. Στην πραγματικότητα, αυτό που φαίνεται σημαντικό είναι ότι το θέμα των 8 ημερών θα μπορούσε να τεθεί στην ελβετική νομολογία. τα πλαίσια εφαρμογής παροχής υπηρεσιών, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την ελβετική νομολογία να το εξετάσει. Αλλά το θέμα που τίθεται είναι η ομοιογενής ερμηνεία των διατάξεων της συμφωνίας που διαθέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συμφωνία λοιπόν, στο άρθρο 16, που προβλέπει την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λέει ότι οι ελβετικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την ομολογία η οποία υπάρχει μέχρι τη στιγμή της υπογραφής. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε καινούριο προκύψει ως νομολογία, κοινοποιείται στις ελβετικές αρχές και το εξετάζει η Μικτή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν μερικώς την εγγύηση της ομοιογένειας. Το θέμα λοιπόν που τίθεται είναι αυτό το ζήτημα της αναλογικότητας του μέτρου άπαξ και πάει στην ομολογία. Η ελβετική νομολογία θα λάβει υπόψη τα κριτήρια τα οποία αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η υποχρέωση έχει να κάνει με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μόνο πριν από το 1999. Έχουμε όμως πολλά παραδείγματα αποφάσεων του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Ελβετίας που λαμβάνει υπόψη αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από την υπογραφή της συμφωνίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι στο βάθος αυτά τα κριτήρια, αυτές οι έννοιες που έχει ερμηνεύσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην πραγματικότητα, ακόμα κι αν υπάρχει περιορισμό στο θεσμικό σύστημα, λαμβάνονται υπόψη εφόσον το επιθυμεί ο δικαστής ο οποίος αναλαμβάνει την υπόθεση αυτή στην Ελβετία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, για να παραμείνουμε στην ελεύθερη κυκλοφορία, υπάρχει μία απόφαση που έχει να κάνει με την νόμιμη παρανομή ενός υπηκό τρίτης χώρας σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομολογία αυτή ακρίς είναι του 2003, μετά δηλαδή την υπογραφή της συμφωνίας το Ομοσπονδιακό Ελβετικό Δικαστήριο τη δέχτηκε. Και πέρυσι, το Σεπτέμβριο δηλαδή πέρυσι, το Δεκέμβριο, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δέχτηκε την ομολογία Μεντόκ επίσης, που είναι το 2008 και που αποτελεί μια αλλαγή στην ε, νομολογία την μέχρι τότε του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το σύστημα λοιπόν έχει τους περιορισμούς του, αλλά την ευθύνη τελικά του δικαστή, μην την ξεχνάμε, αυτός ο Ελβετός δικαστής θέλησε να ε, φροντίσει για την εκπαραλλήλου εξέλιξη της νομολογίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας, παρόλο που δεν είχε την υποχρέωση. Προσπάθησε να το κάνει. Είναι ανοιχτό το ζήτημα. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε κατά πόσο τα κριτήρια της νομολογίας για την αναλογικότητα και τα συνοδευτικά μέτρα θα βρουν σύμφωνους τους ελβετικούς δικαστές ή όχι. Αλλά το σύστημα εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο που δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν ξέρω αν ήμουν αρκετά ξεκάθαρη. Υπήρχε και μια άλλη ερώτηση για την εξέλιξη του θεσμικού συστήματος, αλλά αν θέλετε πρόεδρε, τη συζητάμε αργότερα. Ναι, αργότερα, γιατί θα ήθελα να ακούσω και τους επόμενους θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα. Σας ευχαριστούμε πάντως. Μας εξηγήσατε κάπως την περιπλοκότητα του συστήματος. Για εμά που δεν είμαστε νομικοί, είναι πολύ χρήσιμο. Αυτά που ακούμε σήμερα το πρωί είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και αποκαλυπτικά για μας. Ο κύριο Βίτ, λοιπόν θα απαντήσει σε κάποιες ερωτήσει που του έθεσε ο κύριο Βαμπ, αν δεν απατώμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Ευρωβουλευτή. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να θέσω την προβληματική της υπόθεσης κασίστης της ζών στην εμπορική της διάσταση. Η Ελβετία, 80% των ε, εισαγωγών έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ένας πολύ μεγάλος εμπορικός εταίρος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δεύτερος μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια λοιπόν που δεν είμαστε μέλη, υπάρχουν νομικές διαφορές που παραμένουν. Ε, ο στόχος των πολιτικών είναι να βρούνε τον τρόπο να μην κολλάμε σε αυτά τα κολλήματα όταν τίθεται θέμα κυριαρχίας, αλλά να βρίσκουμε πρακτικούς τρόπους για να λειτουργεί η αγορά και οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των χωρών μας. Αυτός και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, θέλαμε να εισάγουμε την αρχή του κασίστη στη ζώνη στην Ελβετία. Να βρούμε δηλαδή ένα ρεαλιστικό τρόπο να ανταποκριθούμε και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν όσον αφορά το εμπόριο ανάμεσα στην Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και μονομερό ελήφθη το μέτρο, γιατί όπω το εξήγησε και η καθηγήτρια, εμείς δεν είμαστε μέλη, καθηγήτρια δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε την αμοιβαιότητα όσον αφορά την υπόθεση αυτή, αλλά Προσπαθήσαμε, αυτό πιστεύω περιμένουν από εμά και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, να είμαστε νομικά δημιουργικοί, ώστε να βρούμε έναν τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα αμοιβαιότητας. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε, μια που δεχόμαστε τα κριτήρια εθνικής παραγωγής και από τις 27 χώρες, είναι μια πρώτη, ε. τα δικά τους κριτήρια παραγωγής αναγνωρίζονται στην Ελβετία. Θέλουμε όμως οι εξαγωγοί μας να μην βρεθούν στην κατάσταση όπου τα προϊόντα τους ξαφνικά δεν μπορούν να προχωρήσουν εξαιτία εθνικών μέτρων που δεν έχουν εναρμονιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι νομίζω απόλυτα θεμητό από την πλευρά μας στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης που έχουμε. Η εισαγωγή λοιπόν μονομερός της, ε, των προδιαγραφών κασίστης της ζών είναι μια πρωτιά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Αν προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο θα πέσουν οι τιμές. Η κατάσταση σήμερα είναι εξή. Η Ελβετία πρέπει να έχει δύο γραμμές παραγωγής. Εκείνη που εξάγει για καθαρά τεχνικούς λόγους, όχι για λόγους ασφάλειας του προϊόντος, αλλά για να τηρούμε τις εθνικές νομοθεσίες στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, πρέπει να προσδιαριστεί το βάρος ενός σαβού διαφορετικά ανάλογα με το αν εξάγεται προς την, Ελβετία, ε, συγγνώμη, προς την Αυστρία ή προς τη Γερμανία. Το ίδιο και για τα μακαρόνια. Λοιπόν, για μια μικρή επιχείρηση είναι δύσκολο. Η Ελβετία έχει μικρές επιχειρήσεις. Οπότε αναγκάζονται να έχουμε δύο γραμμές παραγωγής, δύο ε, διαφορετικούς τρόπους παραγωγής, ανάλογα με το προς τα που εξάγουμε το προϊόν μας. Το κόστος καταλαβαίνετε ότι είναι περιττό. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την τολμηρή πολιτική χειρονομία. Να πούμε, έχουμε εμπιστοσύνη στους εθνικούς κανόνες. Εννοείται η Κομισιόν του ελέγχει βεβαίως και οι αρχές των κρατών μελών. Δεχόμαστε να τους σεβαστούμε. Είναι θεμητό από την άλλη στη συμφωνία που έχουμε σήμερα στον τομέα των αγροτικών προϊόντων να υπάρξει και κάποια κατανόηση Ακόμα και αν νομικά δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίσουμε την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχει όμως τρόπος να το κάνουμε αυτό διαφορετικά. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σήμερα στους συναδέρφους μας που διαπραγματεύονται με εμά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να βοηθήσουν την εταιρική αυτή σχέση που είναι εξαίρετη σε εμπορικό επίπεδο και από την οποία υποφελείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε ένα ισοζύγιο εμπορικό θετικό όσον αφορά τις εμπορικές σας σχέσεις μαζί μας. Ας βρούμε λοιπόν μαζί αυτά τα μέσα. Να, ποιο είναι το μήνυμα που σας μεταφέρω σήμερα, συμπυκνωμένο. Πρόεδρος, αργότερα ίσως ε, καθηγήτρια Τσούλη, να πάρετε το λόγο. Έτσι καλώς θα είσαστε στο πάνελ μετά, οπότε μπορείτε να απαντήσετε μετά αν δεν σας πειράζει αν δεν έχετε κάτι πολύ δικό να πείτε τώρα. Γιατί θα ήθελα να περάσουμε στις επόμενες δύο παρουσιάσεις και μετά να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Συνεπώς, συνεχίζουμε τώρα και περνάω σε θέματα που έχουν να κάνουν με δημόσιες προμήθειες, που είναι πολύ κεντρικό θέμα στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι που έχουμε εδώ τον Στίβεν Θερχούλστ που είναι εδώ από την εποπτική αρχή των χωρών ΕΖΕΣ και ασχολείται με το θέμα των δημοσίων προμηθειών. Χαίρομαι επίσης που έχω εδώ και τον κύριο Άουντον Σκέιτσφολ, δεν ξέρω αν προφέρω καλά το όνομά σας, που είναι από το Νορβηγικό Συμβούλιο του Καταναλωτή. Για 10 λεπτά θα δώσω το λόγο στον κύριο Φελχούστο όμως πρώτα και μετά σε εσά κύριε Σκέιτσφολ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Εποπτικής Αρχής ΕΖΕΣ θέλω να σας εκφράσω την ικανοποίησή μου που μας δίνετε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ και να σας εξηγήσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δουλειά μας. Έτσι μας γνωρίζετε καλύτερα. μου ζητήσατε να πω δύο λόγια για την πολιτική μας, εποπτεύοντας την εφαρμογή και την θέση σε ισχύ των κανόνων δημοσίων προμηθειών στις χώρες ΕΟΧ. Πριν περάσω στην ουσία του ζητήματος, όμως, θα ήθελα να επενθυμίσω προκαταρτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Διότι εφόσον πράξεις εγκρίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που ξεκινάει πριν οι πράξεις αυτές να φτάσουν στις χώρες ΕΟΧ. Αυτό σημαίνει ότι άπαξ και εγκρίνεται μια τέτοια πράξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά ακολουθείται μια διαδικασία στις χώρες ΕΟΧ που την εξετάζουν, να δουν αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, να δουν μήπως πρέπει να γίνουν συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά λαμβάνεται και απόφαση από την Μικτή Επιτροπή η οποία έχει εκπροσώπους και από τις χώρες ε, ΕΟΧ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς υπάρχει ένα παράλληλο σύστημα, υπάρχουν δηλαδή παράλληλοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες ΕΟΧ. Όμως η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές στην καθημερινή μας δουλειά παρατηρούμε και στις ευρωπαϊκές χώρες καθυστερήσεις. Θέλω να έρθω τώρα στο τελευταίο πακέτο, την ε, οδηγία που την τελευταία που καθορίζει την κατάσταση όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Είναι δύο οδηγίες οι οποίες εγκρίθηκαν το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέθηκαν σε ισχύ το 2006 μόνο. Οι οδηγίες αυτές εγκρίθηκαν στο σύστημα ΕΟΧ το 2007 και τέθηκαν σε ισχύ το 2007. Και μάλιστα το Λίχνενστάιν προχώρησε στη θέση σε ισχύ το 2008. Βλέπετε λοιπόν τις καθυστερήσεις που προκύπτουν εξαιτία της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες σε όχο. Γενικά μιλώντας πάντως μπορώ να σας πω ότι το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες που έχει να κάνει με 10 βασικά πράξεις. Αυτό εφαρμόζεται και στις χώρες ΕΟΧ. Περιμένουμε τώρα να συμπεριληφθούν ε, και οι νέες οδηγίες και περιμένω ότι αυτό θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε σε εφαρμογή το Δεκέμβριο του 2009. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες διαφορές. Κατόπιν τούτου θα σας εξηγήσω ποια είναι η δικιά μας η πολιτική. Πώς εποπτεύουμε εμείς την ε, εφαρμογή και τη θέση σε ισχύ των ε, πράξεων αυτών. Θα έλεγα ότι είμαστε σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ε, πολιτική μας εποπτείας όσον αφορά την εφαρμογή των ε, πράξεων, ΕΟΧ, και μετά έχουμε και εσωτερικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των οδηγιών και των συστάσεων στις χώρες ΕΟΧ ΕΖΕΣ. Όσον αφορά τις οδηγίες, οι χώρες ΕΖΕΣ είναι υποχρεωμένες να μας στείλουν κοινοποίηση της εφαρμογής και στη διαδικασία αυτή ζητάμε από τις χώρες ΕΖΕΣ να μας προμηθεύσουν και ε, τα σημεία αναφοράς, αντίγραφο του νομοθετικού κειμένου και μετάφραση στα αγγλικά ή δυνατόν. Μερικές φορές ετοιμάζουμε και κάποιους πίνακες αντιστοιχιών που στέλνουμε στις χώρες ΕΖΕΣ. βάσει μάλλον του πόσο περίπλοκο είναι το θέμα και το πόσο σημαντική είναι η πράξη, μπορεί να κάνουμε και μια αξιολόγηση συμμόρφωσης με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και όταν πρόκειται για κανονισμούς. Το σύστημα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, όπου εφόσον τρεις μήνες μετά τη συμμόρφωση δεν έχουμε επιβεβαίωση της εφαρμογής ξεκινάμε τις διαδικασίες προσφυγής, επί παραβάση δηλαδή, ε, μετά αιτιολογημένη γνώμη και μετά σε ένα χρόνο εφόσον δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση φτάνει το πράγμα ε, στην ρυθμιστική αρχή στο δικαστήριο. Καταλαβαίνετε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε προσπαθήσει να είμαστε αυστηροί με το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σκέλος της πολιτικής μας και έχουμε στο δεύτερο σκέλος που είναι οι προσφυγές, οι ίδιες πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε σε περίπτωση δημοσίων ε, προμηθειών. Για να σας δώσω μια ιδέα, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ξεκινήσει 8 διαδικασίες προσφυγής με ίδιες πρωτοβουλίες έρευνας. Υπό το φως αυτών, μπορώ επίσης να σας πω ότι εκτιμώντας τις περιπτώσεις αυτές, δεν κοιτάμε μόνο τις πράξεις που εφαρμόζονται στον ΕΟΧ, αλλά εξετάζουμε και ερμηνευτικά κείμενα, τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξετάζουμε ανακοινώσει. Είναι και αυτά μέσα ήπιου δίκαιου που χρησιμοποιούμε εμείς στη δουλειά μας. Εγώ προσωπικά συμμετέχω και σε συμβουλευτικές επιτροπές. Προσπαθούμε δηλαδή να παρακολουθήσουμε πολύ κοντά τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανάλογα να προχωρήσουμε στη δικιά μας τη δουλειά. Όσον αφορά την πολιτική μας λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις προσφυγής, ίδιας πρωτοβουλίας, και εδώ μιλάω για συγκεκριμένες συμβάσεις, συγκεκριμένες διαδικασίες που εξετάζουμε. Παραδοσιακά έχουμε κάποια ιδιαίτερη πολιτική. Δηλαδή, έχουμε μια πρώτη αξιολόγηση. Αν το συμπέρασμά μας εκεί είναι ότι υπάρχει παράβαση των κανόνων ΕΟΧ, τότε στέλνουμε επιστολή στις χώρες ΕΖΕΣ εξηγώντα τα ευρήματά μας και δίνουμε την ευκαιρία στις χώρες ΕΖΕΣ να αναγνωρίσουν, να συμφωνήσουν με τα δικά μας τα συμπεράσματα και μετά να προχωρήσουν σε δήλωση που να λέει ότι θα φροντίσουν οι αρμόδιες αρχές δεν θα κάνουν άλλη φορά τέτοιου είδους παραβάσεις. Αν έχουμε αυτή τη δήλωση, αυτή την αναγνώριση από τις χώρες ΕΖΕΣ, κλείνουμε την υπόθεση. Ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι ότι αυτό είναι συμβατό με την γενικότερη ιδέα που έχουμε ότι το να ζητάμε αποζημιώσεις είναι θέμα εθνικό. Και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να χρησιμοποιούν τις εθνικές διαδικασίες από αυτού. Επίσης ένας άλλος λόγος ήταν ε, πρακτικός. Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις στον τομέα των δημοσίων προμηθειών Και οι χώρες εσές έχουν και τις δικές τους διαδικασίες προσφυγής. Με τη διαδικασία αυτή που ακολουθήσαμε περιορίστηκαν οι προσφυγές που έφταναν σε εμά. Τώρα βέβαια αναθεωρούμε κάπως την πολιτική μας και προσπαθούμε να είμαστε πιο αυστηροί, κυρίως με διάφορους τύπους συμβάσεων. Μακροπρόθεσμα ή όπου διακυδεύονται πολύ μεγάλα ποσά. Εξαιτίας πρόσφατων ε, περιπτώσεων που εξέτασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που δίνει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγκάσει τα κράτη-μέλη που έχουν ε, κάποια παράβαση σε εθνικό επίπεδο να διακανονίσουν την παράβαση αυτή. οι συζητήσεις που γίνονται στο εσωτερικό μας συνεχίζονται. Δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Τελειώνουν όπου να είναι. Οπότε θα σταματήσω εδώ την παρουσίασή μου, ελπίζοντα ότι σας έδωσα να καταλάβετε λιγάκι τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Well, thank um, Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Φερχόλστερ. Χαιρόμαστε γιατί τα μέτρα που παίρνετε είναι αποτελεσματικά και έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Και και ε, ε, βλέπω ότι όλοι οι υπεύθυνοι και από την Κομισιόν και από τα, τα μέλη της Επιτροπής ε, συγκατανεύουν έτσι θετικά, ε, συγκατένευαν μάλλον όσο μιλούσατε. Τώρα θα δώσω λόγο στον κύριο Άουντουν Σκάιτσβολ και ελπίζω να μην δολοφονώ το όνομά σας, λέει ο Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, όπως και αν λέγεστε και όπως και αν προφέρετε το όνομά σας, σας καλωσορίζουμε ιδιαιτέρως ε, στην ε, σημερινή μας συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Ε, και να πούμε ότι ε, στις 15 Μαρτίου στη Μαδρίτη συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα και θα προσπαθήσω να σας ε, πω πώς τα βλέπει και η ΕΦΤΑ. Να σας πω δύο λόγια όσον αφορά το υπόβαθρο. Ήδη ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα αυτό το 2004 όσον αφορά ε, το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο των ε, συμβάσεων. Βασιστήκαμε δηλαδή σε αυτή την έρευνα για αυτό το, το δίκαιο και βασιστήκαμε επίσης και στην πρόταση του Νοεμβρίου 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την διαρκώς μειούμενη κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, βασιστήκαμε επίσης ε, στο γεγονός ε, ότι στην Ευρωπαϊκή Πρόταση γινόταν αναφορά για την μείωση των δικαιωμάτων προς εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών και ευρύτερης επιλογής. Εμείς θεωρήσαμε ότι η πρόταση ενδεχομένως ε, έδινε υπερβολική σημασία στο εμπόριο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 70% του κοινού φαίνεται ότι δεν έχει αγοράσει ποτέ κάτι διασυνοριακά ε, στο ίντερνετ. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στις χώρες ε, ΕΖΕΣ. Φαίνεται ότι το αντίστοιχο νούμερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 12%. Απ' την άλλη πλευρά, είναι σοφή η προσπάθεια να ε, δούμε πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά το διαδίκτυο και τις αγορές ε, online. Εμείς ε, κάναμε αρκετή έρευνα, εμείς οι ίδιοι όσον αφορά το θέμα αυτό και μάλιστα την ξεκινήσαμε ήδη από το 2007. Κάναμε λοιπόν μια ενδελεχή έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ε, είδαμε ότι 45% των καταναλωτών έχουν ήδη ε, αγοράσει κάτι δια της ηλεκτρονικής οδού στο εξωτερικό, ενώ η εθνική διείσδυση είναι της τάξης του 98%. Επίσης, είδαμε ότι είναι δύο τα κυρίαρχα προϊόντα, δηλαδή τα εισιτήρια ε, και τα ταξίδια, ε, αλλά και η αγορά προϊόντων από δεύτερο χέρι, μεταχειρισμένων προϊόντων. Ένα άλλο έβριμα ήταν ότι ο λόγος για τον οποίο πολλοί δεν επιλέγουν την ε, διασυνοριακή συναλλαγή ε, είναι ότι υπάρχει χαμηλή προστασία καταναλωτών κατά 61% ε, και ελλειπής ασφάλεια κατά 60%. Και επίσης ε, ε, είδαμε βάσει της έρευνας ότι οι καταναλωτές δεν ελέγχουν συνήθως τους όρους ε, της σύμβασης. Από πλευράς τώρα πολιτών δεν είδαμε σαν μέρος της έρευνας ότι οι εθνικές, ε, οι διαφορές δηλαδή μεταξύ των εθνικών διατάξεων ε, αποτελούν σημαντικό πρόσκομα στο διασυνοριακό εμπόριο. Όμως ε, δεν θα εκπλαγείτε εάν σας πω ότι ε, καταλήξαμε όσον αφορά την προστασία των, ε, των, ε, την προστασία των ιδιωτικών προσωπικών δεδομένων και της προσωπικής ζωής, καταλήξαμε σε ένα νέο όρο που τον ονομάζουμε contract apathy. Δηλαδή ότι οι καταναλωτές στην ουσία δεν βλέπουν τους όρους της κάθε σύμβασης, αντίθετα από αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πιστεύουμε. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ασφαλές το περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου για τους ε, ε, καταναλωτές έτσι ώστε να, τον να θεωρήσουν το διαδίκτυο ένα συνήθι χώρο συναλλαγών. Επίσης ε, θελήσαμε να μειώσουμε τον χρόνο για την υποβολή παραπώνων ή αντιθέσεων. Ξέρετε ότι μέχρι τώρα φτάνει σε, από δύο σε πέντε χρόνια στην Ορβηγία Επίσης δίνεται στον πολιτή ε, ένα νέο δικαίωμα 37 ημερών ε, για την ακύρωση της ε, σύμβασης και επίσης μειώνει την δυνατότητα να θεωρηθούν άδικη η όροι της ε, σύμβασης. Εμείς πιστεύουμε ότι η προστασία των ε, δικαιωμάτων των πολιτών, των καταναλωτών ε, πρέπει να ενδυναμωθεί και αυτή είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Επίσης θα πρέπει να τους προστατέψουμε τους καταναλωτές από προϊόντα τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί σωστά, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας, ασφάλειας κτλ και βεβαίως ε, θέλουμε ε, και για τις αγορές ε, online να υπάρχει συνολική προστασία. ικανή προστασία και όσον αφορά τις αγορές και όσον αφορά τις πληρωμές. And we also think that you should have additional tools for consumer redress. Um, Τέλος, όσον αφορά την ε, εναρμόνιση, πιστεύουμε ότι η εναρμόνιση θα πρέπει να γίνει στο μέγιστο βαθμό ε, μονάχα όμως οπουδήποτε η έλλειψη εναρμόνισης προκαλεί προσκόμματα προς το ελεύθερο εμπόριο. Μελέτησα λίγο το θέμα αυτό και ε, νομίζω ότι θα πρέπει να το μελετήσουμε περαιτέρω. Εναρμόνιση λοιπόν, η εναρμόνιση αξίζει εάν ε, βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Και βεβαίως θέλουμε και για το μέλλον ε, ε, κανόνες εναρμονισμένους που θα είναι σαφείς, που θα είναι συγκεκριμένοι και που δεν θα πρέπει να αναδιαμορφώνονται κάθε τόσο. Βεβαίω πρέπει να σα πω ότι οι χώρε ΕΖΕΣ έχουν κοινού στόχου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουν αυξημένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καθώ επίση και σοβαρή ε, και αξιόπιστη επιχειρηματική πρακτική. Και νομίζω ότι εδώ είναι ένα καλό σημείο για να τα σταματήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο εισηγητής ε, για θέματα προστασίας των καταναλωτών ε, βρίσκεται εδώ μεταξύ μας, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα μπορούσατε να συζητήσετε εκτός, ε, των, εκτός της θούσης. Μπορείτε να φάτε μαζί για να συζητήσετε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Θα βρείτε πολλά κοινά στοιχεία. Ωραία λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις πριν προχωρήσουμε στο τρίτο τμήμα, το τρίτο σκέλος μάλλον του πάνελ μας. Ε, υπάρχει άραγε κάποιο συνάδελφος ο οποίος θέλει να υποβάλει κάποιο ερώτημα σε σχέση με τις δύο τελευταίες παρουσιάσεις που ακούσαμε όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Α, βλέπω μεταξύ μας ε, τον κύριο Ρούμπιχ ο οποίος ε, ε, είναι μέλος της αντιπροσωπείας με την Ελβετία και τις υπόλοιπες χώρες ΕΖΕΣ. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί εκπροσωπεί το θεσμιθετημένο διάλογο του Κοινοβουλίου με τις χώρες αυτές. Ο κύριος Σβάμπ θέλει να υποβάλει ερώτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φερχούλστ και τον κύριο Σχάιτσφολ για τις ε, παρουσιάσεις τους και να πω ότι, να τους ε, διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις. Ούτως ή άλλως η αλλως η που μόλις έφυγε κάνει μια έκθεση για, την, για τις δημόσιες προμήθειες Φαντάζομαι ότι θα σας ενδιαφέρει και σας και μας είναι ε, σημαντικό για μας να υπάρχει έτσι ένα ίσο, ένας ε, ισότιμος θεμητός ανταγωνισμός γιατί υπάρχουν και οι σχέσεις μας με την, ε, με την Κίνα. Πολλές ε, κινέζικες εταιρείες έρχονται εδώ, εγκαθίστανται στην Ευρώπη, μπαίνουν στην ιστορική αγορά και μετά με κρατικές επιχορηγήσεις δημιουργούν προβλήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω και πάλι την ε, καθηγήτρια Τόμπλερ. Κατά την άποψή σας, η αναλογικότητα μιας ρύθμισης, κατά πόσο είναι δεδομένη σε ένα συγκεκριμένο ε, για τους ε, εργαζόμενους όταν υπάρχει ήδη προκοινοποίηση της σύμβασης. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Ναι, για την προηγούμενη συνεδρία, για την προηγούμενη παρουσίαση, συγγνώμη, είναι η ερώτησή σας βέβαια. Ευχαριστώ. Για το συγκεκριμένο σημείο. Το παράδειγμα που αναφέρθηκε ήταν η κοινοποίηση των 8 ημερών και το κατά πόσο αυτό είναι αποδεκτό στα πλαίσια του διμερούς ε, δικαίου. Από την νομική πλευρά του πράγματος, σε τέτοιε περιπτώσεις υπάρχει, υπάρχει μια απέτηση η οποία εφαρμόζεται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών εκτός Ελβετίας. Και αυτό είναι η διακριτική μεταχείριση. Είναι ιδιαίτερος προβληματικό. Η Ελβετία έχει προσπαθήσει να πει ότι αυτή η απέτηση καλύπτεται από τη διάταξη που υπάρχει στη διμερή Συμφωνία που αναφέρεται στην νομοθεσία για, την, ε, για τους εργαζόμενους. Για την προστασία δηλαδή της θέσης του εργαζόμενου, των ε, συνθήκων εργασίας, των συνθήκων απασχόλησης. Και αυτό είναι ένα πρώτο τεστ που πρέπει να περάσει. Οπότε αυτή η ε, περίοδος όντως έχει να κάνει με την προστασία των εργαζομένων. Οπότε εφόσον έχει κάτι να κάνει με, έχει σχέση με την, ε, ε, με την προστασία των εργαζομένων πρέπει να υπάρχει και αναλογικότητα. Ίσως να μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο επικριτικοί με βάση και το ότι αυτή η απέτηση δεν ισχύει μόνο στην Ελβετία αλλά και σε άλλες χώρες. Όταν μιλούμε για αναλογικότητα, ένα θέμα ουσία είναι ότι το μέτρο που θα επιλεγεί θα είναι το λιγότερο περιοριστικό. Πρέπει να είναι κάτι που θα είναι απόλυτα απαραίτητο. Αν υπάρχει κάτι που είναι λιγότερο περιοριστικό, αυτό είναι που θα πρέπει να προτιμηθεί. Αν τώρα δούμε την ομοθεσία του δικαστηρίου και τις αποφάσεις για προέγκριση ας πούμε και τις σχετικές απαιτήσει, αν αμφισβήτητα το δικαστήριο θα σας πει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αρκεί μόνο να ενημερώσουμε τις αρχές. Ταυτόχρονα επιτρέπουμε να, να συνεχιστεί και η οικονομική δραστηριότητα χωρίς οποιαδήποτε προσκόμματα ή καθυστερήσεις. Και αυτό δεν συμβαίνει, δεν συμβαίνει εδώ. Δηλαδή θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, συνάδει αυτό με, τις με την αρχή της αναλογικότητας, να λαμβάνονται δηλαδή 8 μέρες για να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Θα μπορούσε να ρωτήσει επίσης κανείς, δεν αρκεί να ζητήσουμε οι αρχές να ενημερώνονται για το πώς παρέχεται αυτή η υπηρεσία και μόλις έχουν αυτή την πληροφόρηση να ελέγξουν αν κάτι δεν πάει καλά ή αν θα πρέπει να αναλυφθούν μέτρα, αντί να μπλοκάρουν καταρχήν για 8 μέρες την ε, δραστηριότητα που αποτελεί μεγάλο πρόσκομα ειδικά για τους μικρούς παροχής υπηρεσιών. Εγώ λοιπόν από την νομική πλευρά του θέματος καθαρά σας λέω ότι είμαι αρκετά αρνητική για το κατά πόσο θα πέρναγε στο, το τεστ ε, του δικαστηρίου εάν έφτανε ποτέ εκεί. Το δικαστήριο είναι όλο και πιο αυστηρό όταν μιλάμε για αναλογικότητα και ειδικά για αυτή την ε, απέτηση του λιγότερου ε, περιοριστικού μέτρου που πρέπει να επιλεγεί. Εάν δηλαδή θέλουμε να προστατεύσουμε τους ε, εργαζόμενους και τις συνθήκες εργασίας τους. Ευχαριστώ. Και στα πλαίσια της οδηγίας για τις υπηρεσίες, αυτό το σημείο ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθιξαν οι μικρές επιχειρήσεις για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Και αυτό ακριβώς θέλει να κάνει η οδηγία αυτή, βάζοντας ε, προϋποθέσεις για τις, ε, για τις ε, αποσπάσεις των εργαζομένων, τις οποίες απέριψε το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν άλλες ρωτήσεις, οπότε ας ακούσουμε τους τελευταίους ομιλητές και μετά θα κάνουμε μια γενική συζήτηση. να δούμε τις μελλοντικέ προοπτικές και τα θεσμικά θέματα. Ο κύριος Ρούμπιχ είναι επισήμως μέλος του πάνελ, οπότε ίσως θα πρέπει να έρθει εδώ μπροστά, αντί να βρίσκεται εκεί στην απομόνωση. Και θα σας παρουσιάσω και τους υπόλοιπους ομιλητές. Η κυρία Τόμπλερ νομίζω ότι θα ξαναπαρέμβει στο τρίτο μέρος της συζήτησης. Αλλιώ μπορεί να θέσει ερωτήσει. Αν έχετε και άλλα σχόλια, ευχαρίστω να σα ακούσουμε. Για τα ερωτήματα θα περιμένουμε την συμβολή σας. Χαίρομαι που είναι εδώ σήμερα μαζί μας η δόκτωρ Ανδρέα Έντνερ Κοχ, διευθύντρια του συντονιστικής μονάδας ε, στο Λίχτενστάιν για, την, ε, για τον ΕΟΧ. Έχει ασχοληθεί και με το Solvit, με το... και ήταν συντονίστρια και του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς. Είναι λοιπόν το σημείο επαφής μας σε ό,τι έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά. Και βεβαίως έχουμε εδώ και τον επικεφαλής τη ε, ελβετικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον πρεσβευτή Ζακ Ντεβάτβιλ. Έχουμε και εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και τον Πολ Ρούμπιχ επίσης. Λοιπόν, τέσσερα λεπτάκια για κάποια εισαγωγικά σχόλια και μετά όποιος θέλει μπορεί να παρέμβει και οι συναδελφοί μου εδώ από το Κοινοβούλιο επίσης έτσι ώστε να έχουμε μια έντονη συζήτηση. Φυσικά δεν περιμένω να μας απαντήσετε στα πάντα σήμερα. Ο εισηγητής νομίζω ότι θα έχει έτσι ένα πλούσιο δείγμα όλων των ιδεών που αναφέρονται στην έκθεσή σας. Λοιπόν, η κυρία Κόχα έχει το λόγο. Πρόεδρε, ε, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ε, δυνατότητα που μου δίνεται να συζητήσουμε τι μελλοντικέ προοπτικές και τα θεσμικά θέματα που αφορούν την εσωτερική αγορά στον ε, χώρο ΕΟΧ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφωνία ΕΟΧ έχει αποδείξει την αξία της για τα τελευταία σχεδόν 16 χρόνια και μετά τη θέση σε ισχύ της ε, συνθήκη τη Λισαβόνα είναι καιρό να, να κοιτάξουμε μπροστά. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ε, στην έκθεση που δίνει πραγματικά μια πάρα πολύ καλή α, γενική εικόνα και κάνει μια καλή περίληψη της λειτουργίας του ΕΟΧ και των α, μελλοντικών προκλήσεων. Θα ήθελα να προχωρήσουμε λοιπόν πέρα από αυτή την έκθεση και να επικεντρωθούμε στις πρακτικές ψυχές της καθημερινής δουλειάς του ΕΟΧ και στους, α, στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Κάποια προκαταρτικά σχόλια για το θεσμικό, τη θεσμική οργάνωση. Η συνθήκη ΕΟΧ ήταν μοναδική και αρκετά ισόρροπη, περιλάμβανε και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα κράτη-μέλη που είναι στην ΕΖΕΣ, την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτερστάιν. Η ιστορική αγορά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σωστά και το ίδιο λειτουργεί σωστά και, η, και ο ΕΟΧ. Ε, το ΕΟΧ ε, οφείλεται στην θεσμική, στο θεσμικό, οργάνωση της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν πραγματικά πολύ δυναμική ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο για την ε, πολιτική ενσωμάτωση. Αυτό φαίνεται από το γεγονό ότι η συμφωνία ΕΟΧ μέχρι στιγμή δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα και έχει καλύψει τι ε, προκλήσει που προέκυψαν από πολλέ αλλαγέ ε, οι οποίε έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1992. Για να, για να μπορέσουμε λοιπόν να πληρώσουμε το στόχο μιας ομοιο, ενός ομοιογενούς ΕΟΧ, τα συμβαλόμενα μέρη πρέπει να εξασφαλίσουν μια κοινή και παράλληλη ανάπτυξη των νομικών καθεστώτων τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στις χώρες ΕΟΧΕΖΕΣ για τομείς που καλύπτονται από την Συμφωνία ΕΟΧ. Αυτό γίνεται ε, με σχεδόν μηνιαίες αποφάσεις από την Μεικτή Επιτροπή και αναφέρεται και στις, ε, στις πράξεις ε, του ΕΟΧ, αστυνομικέ πράξει του ΕΟΧ, που είναι περίπου 6.000. Όλα και τα τρία κράτη τη ΕΟΧ ΕΖΕΣ έχουν δεσμευθεί ότι θα συμβάλλουν ε, για να λειτουργεί καλά η εσωτερική αγορά και αυτό φαίνεται από την εξαιρετική εφαρμογή που έχουμε. Σύμφωνα με την τελευταία, το τελευταίο βαθμολόγιο τη εσωτερική αγορά τη ε, Προπτική Αρχή τη ΕΦΤΑ, το έλλειμμα εφαρμογή στο Λίχτενστάιν είναι 0,4% μόλι, τη Νορβηγία 0,5% και τη Ισλανδία 1,3%. Οι χώρες ΕΟΧΕΖΕΣ ε, επίσης θα επιθυμούν να εξασφαλίσουν μια ομοιόμορφη εφαρμογή του ε, δικαίου για τον ΕΟΧ. Αυτό, ε, για, αυτό, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει εμπλοκή και των εμπειρογνωμόνων από τις χώρες ΕΟΧΕΖΕΣ για να εκπονηθούν νέοι κανόνες. Η δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκές επιτροπές, σε εφαρμοστικά εργαστήρια κλπ από πρακτική πλευρά είναι σημαντικό για την θετική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ομοιόμορφη εφαρμογή και ε, διεκπαιρέωση της εσωτερικής αγοράς και των κανόνων της. Το γεγονός ότι τα κράτη ΕΖΕΣ μέχρι τώρα έπαιρναν μέρος σε περίπου 500 ευρωπαϊκές επιτροπές, πέρα από το ότι είναι το δυναμικό στοιχείο της συμφωνίας ε, ΕΟΧ, είναι ένας από τους βασικούς λόγους γιατί η ομογένεια αυτή ε, θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί και αυτό θα ε, γίνει ακόμη πιο σαφές ε, και στα πλαίσια ε, των παρουσών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα θα μπορούσα να σας πω και κάποια πράγματα για την ε, οδηγία για τις, για τις υπηρεσίες, μια που ήμουν και υπεύθυνη για την εφαρμογή της. Τώρα, ποιες είναι οι βασικοί, οι μελλοντικές προκλήσεις. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιολογήσουμε την εμπλοκή, την σχετικότητα που έχει ο ΕΟΧ με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Παρόλο που οι αλλαγέ αυτέ δεν αλλάζουν άμεσα την ε, συμφωνία ΕΟΧ, μπορεί να, την καταστήσουν πιο, ε, μπορεί να καταστήσουν πιο δύσκολο το να αξιολογήσουμε κατά πόσο, ε, σε ποιο, κατά πόσο είναι σχετικό πλέον ο χώρο ΕΟΧ και σε ποιο βαθμό. η ύπαρξη του ΕΟΧΟ έχει χρησιμοποιηθεί ως δείκτη για το κατά πόσο η νομοθεσία είναι εφαρμόσιμη. Αλλά μάλλον ε, δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε νέα προβλήματα λόγω αυτού, μια που οι μεμονωμένε αξιολογήσει τη σχετικότητα των, σχετικό, των ε, πράξεων ούτω ή άλλω ε, γίνονται. Εμεί, οι τρει χώρε τη ΕΖΕΣ, έχουμε κάνει μια συμφωνία με άλλους για, άλλες, για άλλους τομείς νομοθεσίας που δεν εμπίπτουν στην, στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας ΕΟΧ. Ας πούμε το πρόγραμμα ανταλλαγής εκπομπών. Οι προκλήσεις λοιπόν δεν είναι καινούριε στην, στις χώρες ΕΖΕΣ, ΕΟΧ. Παρ' όλα αυτά η αναφορά στους πυλώνες θα, θα χρειαστεί να μελετηθούν, θα δημιουργήσει την ανάγκη να μελετηθούν νέες πράξεις για να δούμε κατά πόσο είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν νέες πράξεις. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η σωστή λειτουργία τη εσωτερική Αγορα πάντα θα την έχουμε υπόψη μα, μια που είναι ουσιώδου σημασία για όλα τα κράτη της, ε, ε, του ΕΟΧΕΖΕΣ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και βεβαίως ε, προσβλέπουμε στην ενισχυμένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Thank you very much. And uh, also... Ευχαριστώ. Το κείμενο υπάρχει, είναι διαθέσιμο, μιλά πραγματικά για πολλά ενδιαφέροντα θέματα και για, την, και για τις πτυχές της οδηγίας, για τις υπηρεσίες. Πάμε τώρα στον κύριο Ντεβάτερβιλ να μας μιλήσει για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση και που κάνατε τον κόπο να καλέσετε και να ακούσετε εκπροσώπους των χωρών ΕΖΕΣ όσον αφορά τις σχέσεις των χωρών ΕΖΕΣ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά πόσο γνωρίζω συμβαίνει κάτι τέτοιο με αυτόν τον τρόπο. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία σας. Οι σημερινές συζητήσεις καταδεικνύουν την σημασία και την περιπλοκότητα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελβετία. Υπενθυμίζω εδώ ότι είμαστε σε μια κατάσταση αρκετά παράδοξη, γιατί γεωγραφικά η Ελβετία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμικά όμως βρίσκεται εκτός. Δεν είναι καν μέρος του ΕΟΧ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενώ είναι ο δεύτερο εμπορικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τι Ηνωμένε Πολιτείε, αν λάβουμε υπόψη μα το εμπόριο, τι υπηρεσίε και τι επενδύσει. Είναι και ο δεύτερος χώρος για εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε ένα πλεόνασμα 15 δισεκατομμύρια με την Ελβετία κάθε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσης, έχει ένα εκατομμύριο υπηκόους που εργάζονται στην Ελβετία και επιχειρήσεις οι ελβετικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν δουλειά επίσης ε, σε πολλούς Ευρωπαίους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που καθημερινά πηγαίνουν για να δουλέψουν στην Ελβετία και γυρνάνε τα σπίτι τους. Όλα αυτά δείχνουν τις καλές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση ε, τέτοιων σχέσεων εμπορικών, ε, οικονομικών, υπάρχουν ομοθεσίες, ε, το ευρωπαϊκό κεκτημένο που συνδυάζεται με στατικές συμφωνίες, καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά που είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση υπάρχουν και τριβές, υπάρχουν και προβλήματα και νέες προκλήσεις. Συγχρόνως όμως γίνονται τεράστιες προσπάθειες για να λύνονται αυτά τα ζητήματα. Μιλήσαμε πολύ για την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων. Το 2008 υπενθυμίζω ότι κάθε μέρα πάνω από 300 Ευρωπαίοι πήγαιναν να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην Ελβετία. Ενώ προς την αντίθετη κατεύθυνση ήταν 10 Ελβετοί την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ασυμμετρία όσον αφορά τα αποτελέσματα που καταδεικνύει αν μη τι άλλο την ε, ελευθερία που υπάρχει η πρόσβαση στην ελβετική αγορά. Οι υπηρεσίε οι διασυνοριακέ τώρα. Επίση, τα τελευταία πέντε χρόνια υπάρχει τεράστια αύξηση, πάνω από 16% ετησίω. Συνεπώ, οι συμφωνίε αυτέ έχουν στεφθεί με επιτυχία οικονομικά. Πάντα βέβαια μπορούν να γίνουν και άλλε βελτιώσει. Η Ελβετία θέλει να συνεχίσει να εμβαθύνει στις σχέσεις αυτές και να τις αναπτύσσει παρετέρω με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μονομερής ε, αποδοχή της ε, υπόθεσης, ε, της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το κασίς της Διζών είναι κάτι που δείχνει τις προθέσεις μας. Οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει επίσης στον αγροτικό τομέα για μια χώρα που είναι πολύ προστατευτική σε αυτό το θέμα, όπως είναι η Ελβετία, δείχνει τη βούλησή μας να αναπτύξουμε παρετέρω τις σχέσεις μας και να επιτρέψουμε παρετέρω πρόσβαση στις αγορές μας. Στις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή την εποχή υπάρχουν διάφορα ζητήματα στα οποία αντιμετωπίζουμε θεσμικές δυσκολίες. Έχουμε νέες προκλήσεις επίσης, όπως για παράδειγμα πώς με μεγαλύτερο δυναμισμό και πιο συστηματικά θα δεχόμαστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και Όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο όπου θέλουμε να διατηρήσουμε την κυριαρχία εκατέρωθεν και θέλουμε καλή λειτουργία των θεσμών επίσης εκατέρωθεν. Είναι μια πρόκληση που είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα είπε ότι τα ζητήματα αυτά που βρίσκουμε σε πολλές ε, υποθέσεις πρέπει να τα δούμε οριζόντια. Άρα ξεκινάει και πάλι ιδέα για μια συμφωνία πλαίσιο. Είναι μια ιδέα ενδιαφέρουσα που αξίζει να την ε, κοιτάξουμε παρετέρω. Από πλευράς της Ελβετίας πρέπει να σας πω ότι θέλουμε να συνεισφέρουμε ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η καλή λειτουργία τόσο των συμφωνιών μας όσο και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλοί από εμά δεν αντιλαμβανόμεθα σε τι βαθμό ο κόσμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάει για δουλειά στην Ελβετία, όπως είπατε. Και το εμπορικό ισοζύγιο, επίσης έχετε δίκιο. Στον κύριο Όλανφερ θα δώσω τώρα το λόγο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Γενική Διεύθυνση Relax. Σα παρακαλώ λοιπόν εκ μέρου τη Επιτροπή έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και σα ευχαριστώ που με καλέσετε. Ναι, Είμαι όντως από τη Γενική Διεύθυνση Relax στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι επικεφαλής της Μονάδας για τις σχέσεις με την Ελβετία και τις άλλες χώρες ΕΖΕΣ, ε, προκειμένου για την εφαρμογή της ε, Συμφωνίας για την Ουστερική Αγορά. Πού βρισκόμαστε στην Επιτροπή από αυτόν Πρώτον, είναι για μας μεγάλη προτεραιότητα οι σχέσεις μας με τις χώρες ΕΟΧ και την Ελβετία. Είναι γείτονέ μας από κάθε άποψη. Η συμφωνία ΕΟΧ είναι πραγματικά μια συμφωνία με χώρε που είναι σχεδόν μέλη, είναι λίγο πιο έξω από το να είναι μέλη. Από το 1994 είναι τελευταία που έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και έχει οδηγήσει σε αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Δηλαδή διασφαλίζει τη συμμετοχή των χωρών ΕΖΑΣ στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπαν και πολλοί προλαλήσαντες, η συμφωνία έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Πρέπει να πω ότι ο λόγος σε ένα μεγάλο βαθμό για την επιτυχία αυτή είναι οι χώρες ΕΖΕΣ οι ίδιες. Διότι έχουν οικοδομήσει ένα πολύ αξιόπιστο σύστημα δύο πυλώνων που είναι αναγκαίο για να τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία αυτή. Φρόντισαν λοιπόν να ενσωματώσουν το εξελισσόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έχουν επίσης μια αξιόπιστη υπηρεσία εποπτείας και έχουν επίσης και πολύ καλή συνεργασία όταν πρόκειται για την νομολογία. Άρα λοιπόν έχουμε χώρες ΕΖΕΣ που συνεργάζονται πολύ καλά επίσης και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν έχει λειτουργήσει τόσο καλά μέχρι τώρα η συμφωνία αυτή. Ποιες είναι οι προκλήσεις τώρα που έχουμε μπροστά μας. Εννοείται ότι οι διαπραγματεύσεις γίνανε 92 με 94. Τότε επικεντρωνόμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην εσωτερική μας αγορά, στην επίτευξη των τεσσάρων ελευθεριών. Ήταν ε, λοιπόν λογικό ότι και η συμφωνία με τις χώρες όχι επικεντρωνόταν σε αυτά. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεκτημένο της, η νομοθεσία της έχει εξελιχθεί και σε πολλούς άλλους τομείς. Μην ξεχνάμε την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την αστυνομική συνεργασία, δικαστική συνεργασία κλπ. Αυτή λοιπόν είναι σήμερα η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Η συμφωνία είναι περιορισμένη, όπως σας είπα, σε θέματα εσωτερικής αγοράς κυρίως. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι στις τελευταίες διαπραγματεύσεις η Επιτροπή μίλησε με τις χώρες ΕΖΕΣ, όμως τώρα υπάρχουν και άλλοι φορείς και άλλοι εταίροι που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις αυτές μετά από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό θα ληφθεί υπόψη στη Νέα Συμφωνία. Υπάρχει μέλλον. Μπορεί να λειτουργήσει μην ξεχνάμε επίση ότι ήμασταν 12 Εμεί και 7 οι χώρε ΕΖΕΣ όταν έγινε η πρώτη διαπραγμάτευση. Τώρα είναι 27 οι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση και 3 οι χώρες ΕΖΕΣ. Καταλαβαίνετε ότι και από αυτό το γεγονό προκύπτουν πολλέ αλλαγέ. Πάντως μπορεί να λειτουργήσει και με δύο χώρε από πλευρά ΕΖΕΣ. Άρα λοιπόν για μας δεν υπάρχει λόγος στο μέλλον να αλλάξει η συμφωνία. Πιο συγκεκριμένα τώρα για την Αλβετία. Εκεί η προσέγγιση είναι διαφορετική, δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω εγώ τους λόγους. Πάντως υπάρχει μια τομεακή και διμερής προσέγγιση. Έχουμε πετύχει πολλά. Έχουμε τα δύο μεγάλα πακέτα, το ένα και το δύο. Αλλά υπάρχουν και περιορισμοί στο τι μπορούμε να πετύχουμε με αυτήν την τομεακή, κατά δηλαδή, προσέγγιση. χρειάζονται πολλά. Και όχι μόνο, όχι τόσο μάλλον από τη δικιά μας την πλευρά. Υπάρχει περιορισμός, είναι πιο στατική προσέγγιση. Την συμφωνία πρέπει να την επαναδιαπραγματευόμαστε κάθε φορά που υπάρχουν αλλαγές, που εξελίσσεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στους τομείς τους καινούριου συνεργασίας που έχουμε για το REACH, για τα μηναρμονισμένα αγροτικά προϊόντα, ηλεκτρισμός κλπ. Σε όλους αυτούς τους τομείς τίθεται τα οριζόντια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να βρούμε δηλαδή πώς θα αντιμετωπίζουμε την εξέλιξη του ευρωπαϊκού κεκτημένου, την ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κλπ. κλπ. Αυτά είναι θέματα οριζόντια, τα είπε και ο πρέσβη, τα οποία πρέπει με οριζόντιο τρόπο να αντιμετωπίζονται στο μέλλον. Και αυτή είναι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την Ελβετία. Εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Um, I think clearly uh, sets out the context. Όντω, βλέπουμε ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο εργάζεται η Κομισιόν και είναι χρήσιμο να το ξέρουμε. Τώρα ο Πολ Ρουμπίχ να μας, μας μιλήσει για κάποια θέματα τα οποία... με τα οποία ασχολείται η Διεκνοβουλευτική αντιπροσωπεία. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που σήμερα εδώ είμαστε μεταξύ φίλων και που η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια πολύ έτσι, μεμονωμένη διαδικασία. Αν δούμε δηλαδή την ιστορική αγορά, τη δημιουργία της, υπήρξαν πολλά διαφορετικά μοντέλα. Κάθε μοντέλο είχε και προτερήματα και μειονεκτήματα. Από τη μια έχουμε αυτούς που επέλεξαν την ολοκλήρωση, εγώ ως Αυστριακός ανήκω σε αυτούς, αλλά πρέπει να πω ότι και η Σουηδία και η Φιλανδία βρίσκονται στην ομάδα αυτή. Τώρα βέβαια εκ των υστέρων βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αποφασιστική σημασία ήταν ότι εμείς ως πολιτικοί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε απολύτως ολοκληρωμένοι. Βρισκόμαστε στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο, έχουμε δικό μας ε, επίτροπο, έχουμε ε, δικα, ε, μια κυρία δικαστή στο, στο δικαστήριο έχουμε πλήρη ενημέρωση και μπορούμε να συναποφασίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν έχει να κάνει με το μέγεθος μιας χώρας, αλλά από την προσωπικότητα η οποία επιδρά και κάνει πιστική δουλειά. Και αυτό γίνεται και σε επίπεδο υπαλλήλων. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς ειδικού, ειδικευμένου υπαλλήλου που πραγματικά είναι εμπειρογνώμονες στην τομέα τους και μπορούν να εξελίξουν τα πράγματα και βλέπουμε ότι αυτό το μοντέλο της ολοκλήρωσης οδηγεί σε μεγαλύτερη συναπόφαση. Και το μοντέλο αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι από τη μια παραδίδει κάποιος κάτι από τις αρμοδιότητές του, αλλά κερδίζει κιόλα από τις αρμοδιότητες των υπολείπων. Δηλαδή από ένα έθνος κράτος πρέπει να μοιραστεί τι ε, αρμοδιότητέ σου με τα υπόλοιπα κράτη. Αλλά αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί ένα κράτος μέλος ε, συναποφασίζει με τα υπόλοιπα 26 και αυτό έχει να κάνει, έχει μεγάλη επίδραση και, σε, και στην εθνική νομοθεσία γιατί όλοι οι υπουργοί βρίσκονται, έχουν το ίδιο πάτημα, κοιτιούνται στα μάτια και αποφασίζουν. Δεν, ισχύει, δεν υπερισχύει η γνώμη του ενός έναντι του άλλου και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Γιατί παρόλο που εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο μιλούμε 23 γλώσσες και το έχουμε οργανώσει και πολύ καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα κατανόησης. Και το, οι συμφωνίες είναι διαφορετικές από ό,τι σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο συνήθως εκλέγεται ένα ε, κόμμα το οποίο ε, δημιουργεί μετά την κυβέρνηση και δίνει τους προσανατολισμούς, δίνει τις γενικές γραμμές και τις εφαρμόζει, στην, ε, αποφασίζει τις, ε, λαμβάνει τις πολιτικές αποφάσεις. Εδώ όμως εμείς χρειαζόμαστε καταρχήν την Κομισιόν η οποία θα λάβει την πρωτοβουλία να εκπονήσει μια έκθεση να εκπονήσει μια πρόταση. Αυτή η εκπόνηση είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία γιατί ξέρετε ότι πρέπει 27 κράτη-μέλη να μελετήσουν τις, ε, την πρόταση αυτή, να ληφθούν υπόψη οι απόψει του, να μπουν σε ένα πακέτο, να βρεθεί αυτό ο ευρύ συμβιβασμό για να καλύπτουν τα συμφέροντα όλων και μετά γίνεται η, δια, η υπηρεσιακή διαβούλευση και στο τέλος αποφασίζουμε με ομοφωνία. Και αυτό πρέπει να γίνει μέχρι, μέσα στα πλαίσια των, ε, της Επιτροπής. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουν και οι 27 Επιτροπή για να έχουμε αρμονία και σωστές αποφάσεις. Αυτό βέβαια δεν γίνεται πάντα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με του υπουργού των κρατών μελών, τι λένε οι άμεσα εκλεγμένοι ευρωβουλευτέ. Και εμεί βεβαίω έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τι τις ε, αποφάσει. Καθορίζονται τα νομικά δεδομένα και, και τα δύο θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, αν έχουν πλειοψηφία μπορούν να συμφωνήσουν επί τη νομοθεσία. Χρειαζόμαστε λοιπόν τρία θεσμικά όργανα. Και εγώ 14 χρόνια εμπειρία έχω εδώ και τα τρία αυτά όργανα πρέπει να σας πω ότι ε, λειτουργούν ανεξάρτητα. Υπάρχει, εντάξει, υπάρχει πίεση βέβαια από τη μία ή την άλλη πλευρά, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη ελευθερία κινήσεων και ότι οι αποφάσεις όντως λαμβάνονται βάσει των ε, αρμοδιοτήτων που έχει το κάθε θεσμικό όργανο. Κλείνοντας λοιπόν, να αναφέρω και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό, αυτά τα θέματα της, ε, της εσωτερικής αγοράς τα επιτύχαμε. Έχουμε μια αγορά που ε, ε, καλύπτει 500 εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά φυσικά διαπιστώνονται και προβλήματα. Για παράδειγμα, για, το, για την κυκλοφορία των κεφαλαίων. Εδώ η εθνική αρμοδιότητα για τη φορολογία έχει παραμείνει στα, η αρμοδιότητα για τη φορολογία έχει παραμείνει στα κράτη-μέλη. Εμείς εδώ έχουμε σε πολλούς τομείς διπλή φορολόγηση η οποία και σχετικές συμφωνίες που δεν είναι εναρμονισμένες και αυτό φυσικά δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, δημιουργεί κινδύνους και έχουμε και σε θέματα φορολόγησης την ε, αρχή την οποία δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τελικά. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, θέλουμε να, είμαστε, ε, ε, να λειτουργούμε κρυπτό. Νομίζω ότι αυτές είναι πολύ σημαντικές πληροφο... συζητήσεις που πρέπει να γίνουν και βεβαίως έχουμε και το θέμα της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Και έχουμε και τα νέα κρατημέλη τα οποία βρίσκονται στην πόρτα μα. Τι νέε υποψήφιε χώρε, συγγνώμη, που βρίσκονται, στη, περιμένουν στην πόρτα μα και πρέπει να δούμε πώ θα μπορέσουν και αυτέ να ενσωματωθούν, αν ενσωματωθούν στην εσωτερική αγορά. Αυτά από μένα και σα ευχαριστώ. Uh, Εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι που εκπροσωπείτε η αντιπροσωπεία σα εδώ σήμερα, γιατί όντω ε, πρέπει να έχουμε πλήρη ενημέρωση για το θέμα τη εσωτερική αγορά. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που ελπίζω να είναι αυτή η ζωντανή συζήτηση που ήθελα να κάνουμε, να μας πούνε όλοι ποιες πιστεύουν ότι είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά τις ε, σχέσεις που έχουμε με τις υπόλοιπες χώρες και για την εσωτερική αγορά. Ίσως σε 30 δευτερόλεπτα να μπορούσαμε να ακούσουμε κάποιες ε, ιδέες δεν ξέρω αν οι συνάδελφοί μου δηλαδή έχουν ε, οποιοδήποτε ερώτημα να θέσουν ε, πριν στραφούμε στο πάνελ. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα τα οποία είναι αρκετά ρεαλιστικά. Σήμερα ακούσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ της συνεργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Και θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ κάποια προβλήματα και να ρωτήσω εδώ τους εμπειρογνώμονες, τους ειδικούς, αν υπάρχουν δυνατότητες επίλυσής τους. Ε, υπάρχουν προβλήματα για την εφαρμογή των συμφωνιών. Οι εποπτικές αρχές ε, είναι διαφορετικές, ακούσαμε για τα δικαστήρια, ε, παρόλο που τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ε, αποφάσεις, το δικαστήριο επίσης έχει τις δικές του, λαμβάνει τις δικές, του αποφάσεις και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είναι αρκετά ε, επαχθείς οι συμφορίες, οι συμφωνίες, η επικοινωνία είναι δύσκολη με τις χώρες ΕΖΕΣ. Ίσως θα έπρεπε από πιο νωρίς να έχουν εμπλακεί στην όλη συζήτηση έχουν γίνει κάποιε προτάσεις και αυτό το θεωρώ καλό, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη πληροφόρηση για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και καλύτερα το τι γίνεται. Επίσης, δύσκολη είναι η εφαρμογή. Λείπουν ε, οι επίσημες κυρώσει, λείπουν προθεσμίες για την εφαρμογή, λείπουν οι συμφωνίες. Όλα αυτά τα θέματα αν μπορούσαν να βελτιώσουν, να μπορούσαν να λυθούν και να βελτιώσουν τι ε, συμφωνίε που ήδη υπάρχουν, θα ήταν πολύ καλό. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Επίση, οι συμφωνίε πλαίσιο και αυτέ πλαίσια πρέπει και αυτέ να τι ε, συζητήσουμε, πρέπει να επιτεχύνουμε, να βελτιώσουμε τις, ε, την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ ρεαλιστικά και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και αν μπορέσουμε να επιτύχουμε στον τομέα αυτό κάποια πρόοδο, έτσι ώστε ακόμη και αυτές οι συμφωνίες που υπάρχουν να, να εφαρμοστούν καλύτερα, θα μπορούσαμε ίσως να βελτιώσουμε και την αμοιβαιότητα που υπάρχει μεταξύ μας, η οποία δεν νομίζω ότι ε, προχωράει πάρα πολύ καλά. Ήδη έχουμε προβλήματα με τις ε, ποσοστώσεις για το γάλα, ξέρουμε πόσα γάλα παράγει η Ελβετία. Ε, αν δούμε πώς ρυθμίζονται αυτά στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου, αυτό να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα. Οπότε η Κομισιόν είναι πολύ ε, συντηρητική σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση. Εν πάση περιπτώσει θα σταματήσω εδώ. Και θα ήθελα να θέσω αυτά τα ερωτήματα στους ε, ειδικούς μας. Πού θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει περιθώριο βελτίωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ζητήσω από τους προσκεκλημένους μας να δουλέψουν πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, θα πω τώρα με ποια σειρά θα σας ζητήσω να απαντήσετε. Αν θέλετε κι εσείς κάτι. Α, ο εισηγητή μα θέλει να ρωτήσει επίση. κάτι. Ναι, πολύ σύντομα θέλω να ρωτήσω κάτι για τις προοπτικές. Και στον ΕΟΧ και στην Ελβετία. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η συμφωνία για το εμπόριο και για τις υπηρεσίες, δηλαδή πώς βλέπετε τις προοπτικές για το μέλλον μιας τέτοιας συμφωνίας. Ας ξεκινήσω από την καθηγήτρια Τούμπερλ και θα προχωρήσω έτσι με τη σειρά για να καταλήξω στον κύριο Φερχούλστ. Αλλά στον πρέσβη θα δώσω το λόγο τελευταία. Το κοινοβούλιο και την επίπεδη τους ακούσαμε, δεν χρειάζεται. Οπότε, σύντομα, συνοπτικά και ο εισηγητής κρατάει το μολύβι του για να σημειώνει τις απαντήσεις σας. Ποιε πιστεύετε ότι είναι οι κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Παρακαλώ, η το Τούμπελ πρώτα. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσει έχουμε από τον Ευρωβουλευτή Κρότσμαν. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά η άλλη είναι, μήπως το σύστημα είναι τόσο περίπλοκο που δεν είναι αποτελεσματικό. Σύντομα θέλω να απαντήσω με το Υπάρχει εδώ μια ανομαλία. Δηλαδή, έχουμε χρησιμοποιήσει μέρο τη εσωτερική αγορά, έχουμε περισσότερη ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων παρά αγαθών εξαιτία τη συμφωνία Σέγγεν. Ένα άνθρωπο μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα ανάμεσα στην Ελβετία και τα κράτη-μέλη, όχι όμω τα αγαθά τα οποία αυτό φέρει. Ένα πολύ απλό παράδειγμα αυτό. Σα δείχνει ότι δεν είναι λογικό όταν μιλάμε για οικονομική ολοκλήρωση. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Αλλά μέσα σε αυτό το περιορισμένο σύστημα ρωτήσατε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του. Η κύρια πρόκληση αναφέρεται και στα επίσημα έγγραφα της Ελβετίας, όπου λέμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα συνεκτικός τρόπος και καλός τρόπος εφαρμογής αυτών που έχουμε πριν πάμε πιο πέρα. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν προκλήσεις όπου πρέπει να περιμένει κανείς νομολογία για να διευκρινίσει κάποια ζητήματα. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζονται νέες συμφωνίες. Έρχομαι σε αυτά που λέει ο εισηγητής για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Βλέπετε στην Ελβετία υπάρχει μικρή αντιμετώπιση. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι καλή ιδέα, άλλοι πιστεύουν ότι δεν είναι καλή ιδέα. Και πρόσφατα η ίδια κυβέρνηση είπε ότι δεν τίθεται θέμα. Ελπίζω να μην είναι αυτή η τελευταία λέξη τους, αλλά καταλαβαίνετε, ακούμε πολλά και διαφορετικά. Πώς τώρα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα. Ε, αυτή είναι πρόκληση και πρόκληση είναι γιατί έχει να κάνει με διάφορα επίπεδα. Δικαστήρια, αρχές, πολιτικούς, ε, διάφορες ενότητες. Εγώ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει μια απλή και εύκολη απάντηση. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω κάτι πιο συγκεκριμένο, αλλά δεν γίνεται. Είναι αδύνατο να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Πολύ ρεαλιστική εξολόγησή σας, λέει ο Πρόεδρος. Εμάς μας αρέσουν οι προκλήσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, κύριε Ράντμαν, εσεί τι λέτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς εξακολουθούν να κρατάνε το ενδιαφέρον του κόσμου και να φροντίζουν για τη συνειδητοποίηση όλων για τα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν ε, εδώ στη σημερινή συζήτηση. Όντως υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να έρθουν. Εμπόδια τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι η διά μου τελευταία λέξη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, η καθηγήτρια Καντούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με την ε, κατάσταση με την Ελβετία, μπορώ να πω ότι η, συμφωνία ύπαρξη διαφορετικών συμφωνιών δυσκολεύει την επίτευξη ενιαίας συμφωνίας. και βεβαίως εάν δούμε συμφωνίες ε, όπως ας πούμε η συμφωνία των αεροπορικών μεταφορών οπωσδήποτε οι διαφορές είναι μεγάλες σε σχέση με, την, ε, με τις ε, συμφωνίες για την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που μας απασχόλησε σήμερα, οι δυσκολίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η κάθε εμπλεκόμενη χώρα προσπάθησε να διατηρήσει την ε, ε, κυριαρχία της ε, νομοθετικά και θεσμικά. Και γι' αυτό λοιπόν όλα συνηγόρησαν έτσι ώστε να καταλήξουμε σε αυτό το ελιπές εργαλείο της Μικτής Επιτροπής. Όμως η κατάσταση είναι αυτή που είναι και βεβαίως μπορούν να ε, υπάρξουν βελτιώσεις, οι οποίες όμως διαρκώς κοντάφτουν στο θέμα της κυριαρχίας που ανέφερα προηγουμένως. Από τη δικιά μου πλευρά θεωρώ ότι σημαντικό είναι ε, να υπάρξει ανάπτυξη δικαίου από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, από πλευράς διμερούς συμφωνίας, δηλαδή θα πρέπει η προσαρμογή του δικαίου και της νομολογίας να γίνεται παράλληλα και από τις δύο πλευρές και το άλλο ζήτημα, στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ε, ο βουλευτής σας, δηλαδή το ότι ε, είχαμε την αίσθηση ότι υπάρχει ε, βούληση εποπτείας κύρωση σε περίπτωση μη εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτό όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν κανείς θέλει να διατηρήσει την νομοθετική ε, ε, κυριαρχία του. βεβαίω μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση για να βρεθούν τα μέτρα βάσει των οποίων μπορεί να γίνει σταδιακή προσαρμογή ε, της νομολογίας γιατί δεν θα πρέπει να βρίσκεται η, η Επιτροπή μία φορά το χρόνο, θα πρέπει να συζητά πολλέ φορές τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό είναι απολύτως ορθολογικό. Δεν ε, εντάσσονται εδώ καθόλου νέες ιδέες ή νέες αντιλήψεις. Για το θέμα της νομολογίας το ίδιο πρέπει να γίνει. Δηλαδή θα μπορούσαν να υπάρξουν δέσμες ενδεχομένως νομολογίας που μέσα από την Μικτή Επιτροπή ε, θα ελέγχονται έτσι ώστε να ενσωματώνονται στην νομολογία. Και τελευταίο στοιχείο βεβαίως είναι η διευθέτηση των διαφορών. Θα πρέπει εδώ να ακολουθηθούν λύσεις ε, οι οποίες έχουν ακολουθηθεί σε άλλες ε, συμφωνίες, αλλά για την προκείμενη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει επικύρωση και από ε, τα δύο συμβαλόμενα μέρη αφενός, αλλά και ευθυγράμμιση των 27 χωρών και της ε, Ελβετίας ε, για, σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για τις τροποποιήσεις ε, της εν λόγω συμφωνίας. Μιλάμε πάντα για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μας δώσατε πάρα πολλές προκλήσεις για το μέλλον, ανοίξατε πολλές σελίδες για το μέλλον. Ε, σας ευχαριστούμε πάντως για αυτό και βεβαίως θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το θέμα. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως ε, ε, συμφωνώ με, τη, τα μας είπε την ερώτημα. Πρέπει να πω ότι θεώρησα και εγώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίαση της ε, ε, κυρίας Τόμπλερ, κυρίως όσον αφορά την λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. Ε, όλα αυτά τα οποία αναφέρει ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε από στενά τις εξελίξεις ε, όσον αφορά τις υπηρεσίες. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέγει ο κύριος Κλοντ Βίλντ. νομίζω ότι θα ήταν όλα πολύ πιο εύκολο αν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού ε, και βεβαίως δεν λέω ότι από αυτού θα πρέπει να βασίσουμε τη σχέση μας αντιθέτως θα πρέπει να δουλέψουμε στενά ε, γιατί όπως όλα τα όσα υπόθηκαν σήμερα καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε ότι έχουμε κοινό μέλλον ότι βρισκόμαστε σε μια κοινότητα στενά συνδεδεμένη από τη μοίρα μας από τη γεωγραφία μας δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η εξέλιξη των σχέσεων. Αυτό δεν είναι δυνατόν πλέον γιατί το επιθυμούν οι πολίτες μας και γιατί έχουμε μεγάλη συνάφεια. Εμπόδια υπάρχουν κόμματα τύπου θεσμικού, τύπου νομικού, αλλά όλα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν ε, όταν υπάρχει πολιτική βούληση η ρεαλιστική προσέγγιση στην ερώτησή σας τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση όπως παρουσιάζεται σήμερα, μπορώ να πω το εξής. Πρώτον, να βελτιώσουμε τις υφιστάμενες συμφωνίες. Η προσπάθεια γίνεται μέσω της εργασίας των μεικτών επιτροπών. Δεύτερον, πρέπει να αναπτύξουμε νέους τομείς συνεργασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εσωτερική αγορά αναπτύσσεται, εξελίσσεται και επομένως η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να ακολουθείται και από την Ελβετία η οποία θα πρέπει να προσαρμόζεται στην τροποποιημένη κατάσταση. Τρίτον, να ενισχυθεί, να σταθεροποιηθεί η σχέση. Ε, κάποιες δυνατότητες δόθηκαν σήμερα το πρωί. Μια συμφωνία πλαίσιο, εάν γίνει αποδεκτή λύση και από τις δύο πλευρές, θα μπορούσε πραγματικά να ισχύσει Ενδεχομένως επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση, ο ένας ε, να είναι πιο πρόθυμος να ακούσει τον άλλον. Ε, πριν από δύο χρόνια ε, αποφασίστηκε η αντιπροσώπευση στην ε, Βέρνη. Έστω και αν η αντιπροσώπευση αυτή ξεκίνησε πολύ αργά, έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες, τις οποίες θα πρέπει να διερευνήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι αισιόδοξη η άποψή σας ότι οι πολιτικοί μπορούν ή θα μπορούσαν να λύσουν ε, τα προβλήματα. Αλλά σας ευχαριστώ που το είπατε πάντως. Κύριος Δεν έχω και πολλά σχόλια να προσθέσω σε αυτά που ε, υπόθηκαν μέχρι τώρα και σε αυτά που είπα και εγώ ε, πριν από λίγο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εμπλεκόμεθα ενεργά στις ε, συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις και μας απασχολούν πολύ κάποια ζητήματα τα οποία βρίσκονται ήδη επιτάπητος και ξέρετε διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα τα οποία ε, εμείς συζητούμε είναι κατά πολύ παρόμοια με τα προβλήματα που συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι βεβαίως η δουλειά που κάνετε ε, για τις δημόσιες προμήθειες. Τώρα τι μπορείτε να μας πείτε εσείς κύριε Σκάιστβολ ε, όσον αφορά τους καταναλωτές. Πολλά ερωτήματα ετέθησαν, αλλά εγώ πρέπει να πω, πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ επικοδομητική μια ανοιχτή συζήτηση όσον αφορά την πλήρη εναρμόνιση των ε, διατάξεων για την προστασία των καταναλωτών Πιστεύω ότι και οι οικονομολόγοι καθώς επίσης και οι νομικές υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν ε, πάρα πολύ. Για την ώρα μπορώ να πω ότι οι αποφάσεις της Κομισιόν θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει οπωσδήποτε με διάφορους τρόπους να ενθαρρύνουμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές να τολμούν να κάνουν εμπορικές συναλλαγές ε, στο διαδίκτυο και ε, διασυνοριακές ε, αγορές. Θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τις καθημερινές ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών και μέσα σε μια ευρύτερη αγορά πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε καλύτερα τα δικαιώματα των ε, ε, καταναλωτών και ε, πιστεύω ότι εφαρμόζοντα σωστά την εσωτερική αγορά οπωσδήποτε βοηθούμε τους καταναλωτές. Και εμεί θέλουμε η συμφωνία να είναι μια επιτυχία στο μέλλον. Βλέπω μια πρόκληση και έχω δύο επιθυμίε. Πρόκληση. Χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι και οι άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ είναι εξίσου ανοιχτέ προ εμά όπω και εσεί είσαστε. Ποιε είναι οι επιθυμίε μου τώρα. Πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι η η υπηρεσία των εξαγωγών όμως να μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο είναι να φροντίσουμε η συνειδητοποίηση και η αξία της συμφωνίας σε όχο για την εσωτερική αγορά να αναγνωριστεί από όλους ότι υπάρχει αυτή η αξία. Ο πρέσβης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ολοκληρώσω με δύο φράσεις. Δύο ρητά, λέει ο μιλητής. Πρώτον, Μερικές φορές το καλύτερο είναι του καλού. Και εδώ θέλω να ε, συμφωνήσω με αυτά που ακούσαμε πριν για το ότι υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, αλλά όχι τόσο των αγαθών και για τον κανόνα των 8 ημερών επίσης. Κοιτάξτε εδώ, είναι ένα ζήτημα γιατί μιλήσαμε για την αναλογικότητα. Όταν μιλάμε για την αναλογικότητα υπάρχουν τεχνικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και θέματα εκτίμησης. Άρα υπάρχει εδώ μια πολιτική διάσταση και οικονομική βέβαια. Όσον αφορά την Ελβετία συγκεκριμένα, ο κίνδυνος για το κοινωνικό dumping και dumping των μισθών είναι υψηλότερος στην Ελβετία που έχει από τα πιο ψηλά επίπεδα ζωής και μισθών στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει να συγκρίνουμε τα μέτρα που λαμβάνονται με τους κινδύνους που ελοχεύουν. Έπειτα υπάρχει και θέμα πολιτικής αποδοχής. Οι αρχές μας λένε ότι χωρίς συνοδευτικά μέτρα δεν θα είχαμε συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Αν λοιπόν σήμερα ε, θέτουμε σε αφισβήτηση τα συνοδευτικά μέτρα, κινδυνεύει η ίδια η ουσία της συμφωνίας. Και γι' αυτό λέω ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού πολλές φορές. Δηλαδή τελικά τι θέλουμε, μια συμφωνία που να λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα ή θέλουμε να τη θέσουμε σε κίνδυνο. Το δεύτερο είναι οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν. Εδώ συμφωνώ με τον εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και συμφωνώ με πολλά που ακούσαμε εδώ για τις θεσμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Εδώ, επειδή μια προσχώρηση που θέλει όλα τα προβλήματα δεν αποτελεί για μας ε, σύντομα τουλάχιστον μια λύση, χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να προχωρήσουμε διμερώς. Και δεν έρχομαι στο δεύτερο ρητό μου που λέει ότι όταν κάποιος θέλει βρίσκει και τον τρόπο για να το κάνει. Αν λοιπόν οι δύο πλευρές καλή την πίστη και με βούληση μπουν σε αυτό το δρόμο θα βρούμε λύσεις αμοιβαία αποδεκτές. Ευχαριστώ. Uh, Ο κύριος Τρακόφσκι θέλει το λόγο. Ε, θέλετε μήπως ε, και εσείς, ο εκπρόσωπο τη Επιτροπής, να πάρετε λόγο. Όχι, α, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάντω που ήρθατε εδώ και συμμετείχατε. Το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Τρασκόφσκι τώρα, για να μα πει τα συμπεράσματά του και να μα πει και πώ προχωράει η έκθεσή του. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επίσης να μας προτείνετε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και όλους τους συναδέρφους που ήρθαν και συμμετείχαν στην ακρόαση αυτή. Έχουμε πολύ τροφή για σκέψη. Πολλά θέματα αποσαφινίστηκαν. Είμαστε στο στάδιο της τελικής έκθεσης. Τη Δευτέρα θα είναι έτοιμη. Και χάρη στην ακρόαση αυτή, πιστεύω ότι θα μπορέσει να είναι πιο συγκεκριμένη. Φαίνεται ότι πολλά προβλήματα στις σχέσεις μας με τις χώρες ε, ΕΟΧ και Ελβετίας έχουν να κάνουν με δικά μας προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις λοιπόν για τις μελλοντικέ προκλήσεις που θα συζητηθούν στην Επιτροπή μας είναι ακριβώς κάτι τέτοιο. Εσείς βασικά έχετε τέτοια προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόθεσή μου στην έκθεση αυτή δεν είναι να κάνω κηρύγματα ούτε να είμαι πατερναλιστής. Όχι, θέλω τη συμμετοχή σας. Και θυμάμαι πριν από λίγο καιρό όταν δούλευα στο Πολωνικό Δικαστήριο για, ε, συγγνώμη, Υπουργείο για την Ολέα, θυμάμαι ότι ερχόντουσαν κάποιοι κοστομαρισμένοι και ερχόντουσαν και μας λέγανε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο να έχετε κάποιον να έρχεται και να σας δίνει μαθήματα. Θέλω συμμετοχή. Και η ακρόση αυτή δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνουμε. Είσαστε πιο σημαντικοί μας εταίροι και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχετε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από πολλές χώρες μέλη. Αν υπάρχουν προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με θάρρος. Και συμφωνώ. Αυτό που είπε και ο Βολτέρος, ότι δηλαδή το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Συμφωνώ. Υπάρχει όμως περιθώριο βελτίωσης και αυτό το θέλουμε βοηθώντας τους οικονομικούς εταίρους, τους οικονομικούς φορείς εκατέρωθεν. Αν αυτό μπορεί να γίνει, ναι. Αν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, γιατί να μην την κάνουμε. Και τη δικιά σας και τη δικιά μας δηλαδή. Τελειώνοντας, ναι, είναι θέμα υπομονής. Συμφωνώ. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο φιλόδοξος στην ε, έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Uh, Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή μας για το ρόλο κλειδί που έχει παίξει στην ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ και τη γραμματεία της Επιτροπής μας που φρόντισε για την ακρόαση. Ευχαριστώ και όλους τους προσκεκλημένους. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε την επαφή μεταξύ μας. Θα δείτε την έκθεση του Τραυσκόφσκι βέβαια στο διαδίκτυο και μπορείτε να μας στείλετε σχόλια. Θα συζητηθεί σε ανοιχτή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ και όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Χαίρομαι που πολλοί προσκεκλημένοι εδώ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι η Επιτροπή μας λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είσαστε όλοι εταίροι μας. Και όλο αυτό το εγχείρημα πρόθεσης της εσωτερικής αγοράς μας αφορά όλους. Είναι, μια... είναι ένα κοινό εγχείρημα και από τις δύο πλευρές. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ που συμμετέχετε με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Είναι μεγάλη ευθύνη και είναι ευθύνη που αναλαμβάνει με πολύ σοβαρότητα η Επιτροπή μας. Γι' αυτό και θέλουμε τη βοήθειά σας. Είσαστε πολίτες, καταναλωτές, επιχειρήσεις που θέλουν να υποφεληθούν από την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και θέλουμε να τους ακούμε. Η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σήμερα ήταν ιδιαίτερα πλούσια. Ανταλλάξαμε απόψεις, πληροφορίες και έχετε και το αντίγραφο της παρουσίασης της καθήτρια Στόμπλερ. Είναι δουλειά που θα μείνει. Σίγουρα θα μας βοηθήσει στη συζήτησή μας και στο έργο μας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που συμμετείχατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Τώρα να πω στα μέλη της Επιτροπής αυτής, τους Ευρωβουλευτές. Θα ξαναβρεθούμε 7 και 8 Απριλίου. Στις 4.30 όμως θα αρχίσουμε στις 7 του μηνός, γιατί υπάρχει μια έκτακτη ολομέλεια για να ακούσουμε τα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής. Οπότε 4,5 με 8 θα είναι η συνεδρίασή μας στις 7 Απριλίου και 9 με 12,5 στις 8 Απριλίου. Θα τα ξαναπούμε τότε λοιπόν και πάλι σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλό ταξίδι!